ευχαριστώ επίσης ε, τα μέλη του Πολωνικού Κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα τον Αντιπρόεδρο της ε, τον ε, κύριο Πομαίδα, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος της Πολωνικής Βουλής και αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας και τους κυρίους Χάικερ και Γκαρμπόνσκι που είναι μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης της Υπέθρου. Επίσης, τον Χωσέ Λουίς Μαρτίνες Γουγιάρο που είναι ο Υπουργός Γεωργίας της Καστίγια Λαμάντσα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Είχαμε πολλές ευκαιρίες αγαπητοί συνάδελφοι τους τελευταίους ε, μήνες που εμβαθύναμε όλες τις προβληματικές ε, για την ε, ΚΑΠ του μέλλοντος. Τώρα έχουμε μπει στο ψητό. Σήμερα έχουμε την ευθύνη να φτιάξουμε μια κοινή αγροτική πολιτική που να ικανοποιεί τις προσδοκίες των πολιτών μας για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις που ενδιαφέρουν στη σύγχρονη κοινωνία. Προστασία του περιβάλλοντος, τροφιμική ασφάλεια, ευημερία των ζώων, ποιότητα της παραγωγής μας. Σε αυτό το πλαίσιο η ΚΑΠ του μέλλοντος πρέπει να παίξει κεντρικό ρόλο. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την πορεία εξυγχρονισμού της ΚΑΠ όπως ξεκίνησε από το 1992 και που συνεχίστηκε με την Ατζέντα 2000 και τη μεταρρύθμιση Φίσλερ του 2003. Θα πρέπει να εργαστούμε για μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση η οποία θα δώσει αξία στην γεωργία και στην Ήπεθρο για να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, προκλήσεις. Θα πρέπει να έχουμε παραγωγή υπηρεσιών, κοινοφελούς έργου από τους αγρότες ε, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε και τη συνέχεια της γεωργικής δραστηριότητας μέσα στο χρόνο να προωθήσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας, την ενίσχυση και τον, ε, την, ενίσχυση των ε, μέσων ε, σύναψη συμβάσεων που έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, Όπως ε, καταμαρτυρεί η κοινοβουλευτική μας δουλειά, στο έγγραφο Ευρώπη 2020 ζητήσαμε σημαντικές τροποποίησεις και όλο το Κοινοβούλιο είπε ότι η Ευρώπη η οποία θέλει να παίξει καθοδηγητικό ρόλο για τις στρατηγικές που θα πρέπει να αναλυθούν για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, αυτή η Ευρώπη δεν θα πρέπει να απαρνηθεί τις επενδύσεις στον τομέα αυτό όπου χρειάζεται και να τον κόσμο. Βρισκόμαστε εμείς σε μια ιστορική φάση με τη Λισαβόνα η συναπόφαση για τα θέματα γεωργίας προσδίδει σε εμά το Κοινοβούλιο έναν δυναμικό ρόλο στην ομοθετική διαδικασία, μας επιτρέπει να ενισχύσουμε το δημοκρατικό προφίλ των αποφάσεων που θα αναλάβουμε στο μέλλον. Είμαι πεπισμένος ότι η σημερινή ακροασία είναι και η κατάλληλη ευκαιρία για να βαθύνουμε στον προβληματισμό μας και για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την τρέχουσα συζήτηση για τον καθορισμό της μελλοντικής ε, ε, ΚΑΠ και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Ο κύριος Τζορτζ Λάιον έχει το λόγο. George, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπατε και εγώ έχω άγχος ε, για να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ προκαταβολικά τους ε, συναδέλφους ε, που συνεισέφεραν στο έγγραφο που παρουσίασα πριν από δύο εβδομάδες. Η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι μια ουσιαστική πρόκληση για την Επιτροπή μας μέσα στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας. Εμείς έχουμε εξουσία και θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη για την ε, οικοδόμηση μίας νέας ε, ΚΑΠ ικανής ε, να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Λοιπόν, να σας αναφέρω μερικές από αυτές τις προκλήσεις και θα δώσω το λόγο μετά στους υπόλοιπους ομιλητές. Η πρώτη πρόκληση είναι η οικονομική, χρηματοπιστωτική κρίση. και η πίεση η οποία ασκείται από αυτήν την κρίση ούτως ώστε η χρηματοδότηση και τα κονδύλια να είναι ιδιαίτερα περιορισμένα. Δεύτερο είναι η αναγκαιότητα να έχουμε ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών και όλων των γεωργών όπου και αυτοί και αν βρίσκονται. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση. Τρίτο, η παραγωγή που θα πρέπει να αυξηθεί που σύμφωνα με την ΦΑΟ ε, προβλέπεται να υπάρξει πολύ μεγαλύτερη ζήτηση τροφίμων στο μέλλον για να αντιμετωπίσουμε <coughs> τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Βέβαια σήμερα υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Γνωρίζουμε ότι λόγω των κλιματικών αλλαγών υπάρχουν δυσκολίες ε, στην διασφάλιση της αυτάρκειας και λόγω του προβλήματος ε, του νερού ε, και του προβλήματος ενέργεια αλλά και των αρρώσιμων γεών που έχουμε στη διάθεσή μας για την παραγωγή μεγαλύτερων ποσοτήτων. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να χρησιμοποιούμε αδιακρίτως ε, τη γη, αλλά θα πρέπει να της προσδώσουμε μία εφορία στη χρήση. Επίσης, εν ώψη αυτής της πρόκλησης θα πρέπει να έχουμε και μία αηφορία του πυρήνα της πολιτικής μας. Δηλαδή εμείς θα πρέπει να παρέχουμε δημόσια αγαθά, κοινά αγαθά, αλλά προστατεύοντας το περιβάλλον ταυτόχρονα. Αυτή είναι μια άλλη δέσμευση ως προς την ικανότητά μας να ικανοποιήσουμε την μεγαλύτερη ζήτηση. Επίσης ε, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι η ΚΑΠ αποτελεί τμήμα της λύσης ε, των νέων προκλήσεων και όχι τμήμα του προβλήματος. Εμείς ε, θα πρέπει να δώσουμε νέες απαντήσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στα πλαίσια του 2020. Οι κλιματικές αλλαγές, η πράσινη και η φόρα ανάπτυξη. Θα πρέπει λοιπόν να αποδείξουμε εμείς ότι μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα του 2020 και η Γεωργία θα πρέπει να γίνει θεμελιώδες ε, ε, στοιχείο επίλυσης του προβλήματος. Και θα πρέπει να συνεχίσει να εξασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα των ε, Ευρωπαίων γεωργών ενάντια των άλλων μεγάλων ανταγωνιστών του, σε παραδείγμα των Ηνωμένων Αυτό είναι ένα πρώτο και πρωταρχικό ρόλος τη κοινή γεωργική πολιτική, αλλά και θα πρέπει να διατηρηθεί η γεωρική παραγωγή σε ολόκληρη την Ευρώπη. Απαραίτητο όρο και για το μέλλον. Και επίσης πληθώρα προσφοράς σε τρόφιμα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η ε, προστασία των ζώων, τη ευημερία των ζώων. Αυτέ είναι οι προκλήσεις. Ελπίζω οι έξι πραγματογνώμονε να δώσουν τι απαντήσει. για να έχουμε με βάση και το έγγραφο συζήτηση τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τι θέσει μα όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία, σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον George Lyon για την παρουσίασή του και συνεχίζουμε δίνοντα το λόγο αμέσω στον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Τάσο Χανιώτη. Έχετε το λόγο. Τάσο. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ευχαριστώ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να συζητήσουμε κάποια λόγια σχετικά με, την, ε, με τις προοπτικές της κοινωνικής πολιτικής μετά το 2013, προοπτικές τις οποίες ασφαλώς και θα επηρεάσει ο ενισχυμένος ρόλος που καλείται από εδώ και μπρος να διαδραματίσει το Κοινοβούλιο ως προς το μέλλον της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ίσως είναι πρόημο το να δώσουμε συγκεκριμένες προτάσεις τώρα, ωστόσο έχουν ήδη ξεκινήσει, το, έχει ήδη ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος σχετικά με το μέλλον της ε, ΚΑΠ και κινείται λίγο πολύ γύρω από δύο βασικά ζητήματα. Χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική όπως έχει αυτή τη στιγμή και χρειάζονται και οι δύο πυλώνες της ΚΑΠ από τη Γενική Διευθυνσία Ιωρικών ε, φυσικά δεν θα σας εκπλήξει το να σας πω ότι όντως ε, καταφατικά απαντούμε και στα δύο ερωτήματα αυτά. Αυτό που έχει προσπαθήσει να κάνει από τη δεκαετία του 90 και μετά η ΚΑΠ ήταν να εξασφαλίσει την προσαρμογή και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων ε, τη εποχή. Για να δούμε λοιπόν ποιε ήταν οι μεγάλε αυτέ προκλήσει. Χαρακτηρίζονται καταρχά από την ανάγκη ε, για την ε, ΚΑΠ να προσαρμοστεί στι συνδυασμένε στις συνδυασμένες επιπτώσεις των, οικονομικής κρίσης και των κλιματικών αλλαγών μέσα στο πλαίσιο και τους περιοριστικούς όρους των περιορισμένων δημοσιονομικών μας πόρων. Θα ήθελα λοιπόν στη σύντομη παρέμβασή μου να περιοριστώ στους κύριους όρους δηλαδή την οικονομική κρίση και τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής. Πρώτο ερώτημα. Και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απαραίτητοι και σχετικοί με τον προσδορισμό του μέλλοντος της ΚΑΠ, δεδομένης και της μεγάλης ψητικότητας των γεωργικών τιμών ύστερα από την ε, μεγάλη ε, από τη μεγάλη άνοδο των τιμών των ε, τροφίμων και μετά την μεγάλη κρίση είναι υψηλότερο τώρα το κόστος ε, input, δηλαδή το κόστος παραγωγής και βέβαια είναι δύσκολο σε τούτου να διατηρηθούν σχετικά χαμηλά οι τιμές και επιπλέον παράγοντες που δεν μπορεί να γνωριθεί είναι η κλιματική αλλαγή. Εδώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μία πτυχή που αναφέρθηκε ε, πολύ γνωρίτερα, ότι η Διεθνής Οργάνωση Γεωργίας ε, έχει πει ότι θα πρέπει στο μέλλον να αυξηθεί κατά ε, μεγάλο ποσοστό η γεωργική παραγωγή, η παραγωγή τροφίμων, ενώ στα προηγούμενα, ώστε μέχρι τώρα χρόνια έχει αυξηθεί κατά 148%, έχουμε ακόμη μεγάλες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Και οι απαντήσεις που θα δώσουμε, όπως και το γεγονός, ε, η απάντηση που θα δώσουμε πρώτα κατά πόσον οι δύο αυτοί παράγοντες, κλιματική αλλαγή δηλαδή και η οικονομική κρίση έχουν και για το μέλλον της ΧΑΠ ε, συνάφεια θα μας καθοδηγήσει και στις απαντήσεις μας. Αυτό λοιπόν όσοι πιστεύουν ότι έχουν σημασία και οι δύο αυτοί παράγοντες ε, καταλήγουν στο συμπεράσμα ότι οι άμεσες πληρωμές παραμένουν σημαντικές για το μέλλον της ΚΑΠ, για την υποστήριξη του δημόσιου αγαθού. Εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι μακροπρόθεσμα μόνο κλιματική αλλαγή θα έχει κάποια σημασία και συνάφεια, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι άμεσες πληρωμές δεν διαφυλάσσουν κάποιο δημόσιο αγαθό. Η ενίσχυση λοιπόν της προμήθειας ή της προσφοράς του δημοσίου αγαθού από την ΚΑΠ θα αποτελέσει και το κρίσιμο χαρακτηριστικό βεβαίως της προσαρμογής νέας πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα και σε συνδυασμό με την προσπάθεια για προστασία των παραγωγών. Και έτσι είδαμε, εξετάσαμε δηλαδή τη δυνατότητα να συνεργαστεί ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα για να αποφύγουμε τις ε, επιδοτήσεις, τις ενισχύσεις από το δημόσιο ε, τομέα. Όπου ναι, μπορεί να προχωρήσει μια παραγωγή έτσι, χωρίς μια ΚΑΠ δηλαδή, αλλά με χαμηλότερη προστασία και προμήθεια ε, δημόσιου αγαθού, με χειρότερες περιβαλλοντικές συνθήκες. Η παρουσία ύπαρξη της ΚΑΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο όρος ο οποίος έχει διαφυλάξει και την ε, εδαφική ισορροπία αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος στην Ήπειρό μας. Έτσι λοιπόν και για το μέλλον της ΚΑΠ αυτή η ερώτηση προσλαμβάνει διαφορετικές αστάσεις εν ώψη της οικονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει σημαντικές απώλειες οδημάτων για τους γεωργούς της Ευρώπης που το 2008-2009 απόλεσαν όλα τα σορευτικά ε, ωφέλη από τη μεταρρύθμιση από το 1994 και μέχρι σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το να πούμε ότι αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν σχέση με την γεωργική πολιτική και έχουν ελάχιστη σχέση με τις εξελίξεις ως προς τις βασικές, τη βασική λειτουργία των γεωργικών αγορών. Ταυτίζονται όμως, συμπίπτουν καλύτερα με την ε, ε, με το χειρότερο σημείο της κρίσης, ίσως παραδοξολογικά, ίσως ως οξύμορο δηλαδή, αλλά πάντως βλέπουμε ότι η ε, κρίση στα τρόφιμα μπορεί να περιγραφή ως περιγραφή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως περιγραφή της μεγάλης κρίσης στη Γεωργία και ταυτόχρονα της μεγάλης υποπάθμισης του γεωργικού ε, εισοδήματος. Η παράλληλη εξέλιξη και των τριών βασικών ε, αγορών, δηλαδή της γεωργίας, της ενέργειας και των μεταλλουργικών προϊόντων, παρότι η εξέλιξη δεν, ε, είναι, δεν ακολουθεί την ίδια ακριβώς πορεία στους τρεις αυτούς τομείς, οι συμπίες που υφίστανται και οι τρεις τους είναι πάρα πολύ σημαντικοί και ιδιαίτερα βλέπουμε την ανάγκη να διαφυλαχθούν κάποια απαραίτητα ελάχιστα μέτρα προστασίας της αγοράς ως ένα ελάχιστο δίκτυο ασφαλείας και για τα προϊόντα για την ε, γεωργία. Ταυτόχρονα όμω θα πρέπει να συζητήσουμε και τον τρόπο λειτουργία τη αλυσίδα των τροφίμων και το κατά πόσο εάν ένα πιο στοχευμένο δίκτυο ασφαλεία για το εισόδημα ω μέσον διαχείριση τη κρίση θα μπορούσε και να εισαχθεί στη μελλοντική ΚΑΠ ε, αντίστοιχες ε, εξελίξεις φυσικά συνδέονται και με το μελλοντικό σύστημα πληρωμών, σύστημα το οποίο προσφέρει ε, το απαραίτητο δίκτυο ασφαλείας για τις γεωργικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα συμβάλλει και στην ε, προσφορά και διαφύλαξη του δημόσιου αγαθού ως έργο που επιτελεί η γεωργία. Για να μπορέσει λοιπόν αυτό το το σύστημα να εξασφαλίσει τους στόχους του και μετά το 2013 διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα όσα έχουμε ήδη επιτύχει μέχρι σήμερα, απαιτείται να εξεταστούν περαιτέρω προσαρμογές προς ένα πιο εναρμονισμένο επίπεδο υποστήριξης, στήριξης καλύτερα. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε κατανομή μεταξύ των, εμπορικών των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των κρατών μελών με βάση την ιστορική τους παραγωγή. Πρέπει να προχωρήσουμε προς μια σύγκληση και μεταξύ γεωργών αλλά και μεταξύ κρατών μελών. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος θα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις σε σκληρά ερωτήματα και το χρονισμό και τις όρους μετάβασης και το κατά πόσον η διαφύλαξη του εισοδήματο μπορεί να αποτελέσει ένα φυσικό μειονέκτημα στην υπόθεση αυτή και το κατά πόσον μπορούμε να καλύψουμε την ψαλίδα μεταστή του στάτου του ΣΚΒΟ και ενό ε, καταποκοπήν προσδορισμένου ελάχιστου εισοδήματο. Αυτό, ωστόσο, όπω και να το συζητήσουμε, θα πρέπει να ικανοποιεί δύο βασικέ ανάγκε. Καταρχά, τη βασική στήριξη εισοδήματο και δεύτερον, τη βασική στήριξη και προστασία του δημόσιου αγαθού. Το οποίο σημαίνει ότι όποια μέτρα εισάγονται, όπως και πρόσφατα με τις προτεραιότητες για την κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να αποτελούν ταυτόχρονα και μέτρα εφαρμογής της κοινή γεωργικής πολιτικής και της, αναθεώρησή τη, αναθεώρησής της, της μορφής, και να επιτρέψουν τα κράτη-μέλη να συμπληρώσουν με, ένα, με μια εργαλειοθήκη, θα λέγαμε, τα υπόλοιπα μέτρα, τα οποία θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, θα βελτιώνουν το περιβάλλον, του και θα εξασφαλίζουν ε, βιωσιμότητα για τις κοινωνίες των γεωργών τους. Άρα, και με τις άμεσες πληρωμές και με τα υπόλοιπα συμπληρωματικά μέσα της ΚΑΠ πιστεύουμε ότι θα πρέπει στο μέλλον να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το δημόσιο αγαθό για την ευρωπαϊκή γεωργία εξασφαλίζοντας δύο ευρύτερους στόχους. Πρώτον ασφάλεια τροφίμων με την διατήρηση της δυνατότητας παραγωγής ε, μάλλον επιστηστική ασφάλεια, με τη διαφήμιση τη δυνατότητα παραγωγή τη ευρωπαϊκή γεωργία και τη διατήρηση βέβαια των ε, γεωργών, την εφορία των θέσεων εργασία του, αλλά ταυτόχρονα και την προστασία του περιβάλλοντο, ε, το φυσικό περιβάλλον, είτε είναι το οικονομικό. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα ε, και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι ξεκάθαρε ιδέε για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τώρα αρχίζουμε το πρώτο μέρο τη ε, ακρόασή μα και ε, αρχίζουμε δίνοντα το λόγο στου γεωργού και στου εκπρόσωπου τη υπαίθρου. Ζητώ λοιπόν από τον αντιπρόεδρο τη ΚΟΠΑ. parola. Γκέρντε Ορλάιτενερ. Έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρετε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σα παρουσιάσω τι απόψει ε, των Ευρωπαίων Γεωργών για την περαιτέρω εξέλιξη τη ε, ΚΑΠ μετά το 2013. Η ΚΑΠ ε, είναι πιο δυναμική και πιο σύγχρονη από ό,τι ίσω νομίζουμε. Έχει προχωρήσει σε πολύ βαθιές μεταρρυθμίσεις και η Ευρωπαϊκή Γεωργία έχει αποδείξει ότι μπορεί με ευελιξία να προσαρμοστεί στις προδοσδοκίες και τις απαιτήσει της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Δηλαδή έχει, έχει ενισχύσει σημαντικά την ασφάλεια των τροφίμων και την επιστηστική ασφάλεια. Έχει ε, ε, και έχει ήδη τηρήσει και τηρεί, εξακολουθεί και τηρεί πολύ ψηλές προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος και των ζώων. Έχει εισαγάγει μέτρα στον τομέα της ανάπτυξης πέθρου και έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες των αγορών. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε προσαρμοστεί, έχουμε ακολουθήσει ένα πολύ σωστό δρόμο, τον οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε και μετά το 2013, χωρίς όμως ε, να μειώσουμε, να υποβαθμίσουμε την ε, ποιότητα της ε, δουλειάς μας. Έχουμε να κάνουμε 50 εκατομμύρια ανθρώπους που εργάζονται σε μεσαίες και, μικρο, σε, και μικρές επιχειρήσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ο τομέας λοιπόν της γεωργίας ε, είναι εκείνος ο οποίος διαφυλάσσει και την ποικιλία του, της υπαίθρου ο γεωργικός πληθυσμός όπως και ο τουρίστας έχει να συναντήσει επισκεπτόμενο στην υπαίθρο μας μία ένα τοπίο γεμάτο διαφορές, γεμάτο ποικιλία και ένα υγιές ε, τοπίο. Ε, όλα αυτά όμως, το κόστος δηλαδή αυτής, αυτών των θετικών πτυχών, ποιος το έχει επομιστεί. Είναι βέβαια ότι δεν το έχει επιμιστεί ο καταναλωτής, διότι οι τιμές του δεν έχουν, ε, δεν έχουν αυξηθεί από τη δεκαετία του 90. Οι τιμές έχουν ε, αυξηθεί μόνο κατά 49% ενώ οι τιμές παραγωγού έχουν αυξηθεί μόνο κατά 27%. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μπορούμε να έχουμε την δυνατότητα να διαφυλάξουμε και το επίπεδο των τιμών χάρη στη δυνατότητα προσφοράς ε, ενισχύσεων στις πληρωμές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησε με μια μελέτη την οποία έχει αναθέσει την οποία ε, για εν του 2020 τη δυνατότητα να, αποφευθούν, να, να επιφευθούν οι καταστροφικές συνέπειες πιθανών περικοπών σε άμεσες πληρωμέ. και δεν θέλω να παραθέσω εδώ τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης όπου ε, αναφέρεται ότι το να μειωθούν οι άμεσες πληρωμές από τον πρώτο πυλώνα σημαίνει και εντατικοποίηση της χρήση τη γη και ε, σημαντική συμπίεση του εισοδήματος για τους γεωργούς. Μόνο 50% του εισοδήματος, ε, το, το μέσο εισόδημα του Γεωργού αντιστοιχεί μόνο σε ένα 50% του εισοδήματος των λοιπόν τομέων και δύο τρίτα αυτού του εισοδήματος προέρχεται από τις άμεσες πληρωμές, σχεδόν το ένα δεύτερο αυτού του εισοδήματος από τους, ε, τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα και χωρίς αυτά, αυτές τις πληρωμές δεν θα μπορούν οι Γεωργοί να διατηρήσουν την προσφορά που ε, έχουν μέχρι τώρα επιδείξει και για την παραγωγή αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με νέες ε, προκλήσεις για τη γεωργία. Ε, λόγω της ε, κλιματικής αλλαγής υπάρχει κίνδυνος και για την παραγωγή και για την ποιότητα της παραγωγής τροφίμων με κίνδυνο για, ολόκληρη, για όλη τη γη, για όλη την ανθρωπότητα, με σημαντικές διακυμάνσεις αγορές και με σημαντικούς ε, κινδύνους επισητιστικούς. Αυτές λοιπόν οι συνθήκες ε, για την κοινή γεωργική πολιτική τι όρους μπορεί να προσφέρουν για την περίοδο μετά το 2013. Ο πρώτος πυλώνας θα χρειαστεί οπωσδήποτε μια κατάλληλη χρηματοδότηση και θα πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση του πρώτου πυλώνα. Από το 2013 και μετά θα πρέπει να είμαστε θέση να διαφυλάξουμε και να διατηρήσουμε την θέση του Γεωργού και της Γεωργίας την, να ενισχύσουμε τη θέση του γεωργού στην ε, αλυσίδα παραγωγής τροφίμων και να ενισχύσουμε και την ποιότητα, την ασφάλεια δηλαδή των τροφίμων. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να αντισταθμίσουμε την πληθυντικότητα των ε, τροφίμων στις αγορές και τις τις συνέπειες των ε, της κλιματικής αλλαγής. Η Ένωση μας λοιπόν, η ΚΟΠΑ ΚΟΣΕΚΑ, προτείνει τα εξής. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν σταθερές και καλύτερες λειτουργίες ε, των αγορών μέσα από τις αγορές με τα σταθμιστικά μέτρα. Οι κρίση στις διάφορες γεωργικές αλλογές που είδαμε τα τελευταία ε, ένα-δύο χρόνια είδαμε, ε, δείχνουν ότι η πολιτική μόνο περιορισμένος μπορεί να παρέμβει και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Η ΚΟΠΑ και η ΚΟΣΕΚΑ θεωρούν ότι θα πρέπει να λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα μέτρα των αγορών ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για τις γεωργικές αγορές ότι χρειάζονται νέα μέτρα και εμείς συζητούμε αυτή τη στιγμή πρόσθετα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, ενίσχυση δηλαδή των οργανώσεων των παραγωγών, μέτρα τύπου δικτύου ασφαλείας ε, ώστε να αντιμετωπίζεται η απώλεια εισοδήματος και τρίτον φορολογικά μέσα σε εθνικό επίπεδο. Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του, γεωργικού, του γεωργού στην ε, αλυσίδα των τροφίμων με μια σειρά μέτρων, με μια ανταγωνιστική πολιτική η οποία δεν θα εκθέτει τον ε, παραγωγό στην απόλυτη πίεση των μεγάλων, ε, των μεγάλων αλυσίδων φτηνών τροφίμων, αλλά θα εξασφαλίζει μάλλον πιο ισόρροπες σχέσεις, έτσι ώστε να είναι και η αλυσίδα των τροφίμων ασφαλής και η ποιότητα των τροφίμων με μια σαφή καθοδήγηση του καταναλωτή ε, όταν επιλέγει ποιο προϊόν θα αγοράσει. Επίσης χρειαζόμαστε μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργού, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις και προτείνουμε τα εξής μέτρα. Ενίσχυση των ε, μέσων ανταγωνιστικότητας από το δεύτερο πυλώνα, προσαρμογή δηλαδή στις κλιματικές αλλαγές, ε, ε, προσαρμογή, μάλλον ανάπτυξη της αιτικής έρευνας, ε, διατήρηση, διαφύλαξη της βιοπικιλότητας, ε, αηφορία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, διατήρηση και αναδιαμόρφωση του ισχύοντος συστήματος άμεσων πληρωμών και εδώ έχουμε να κάνουμε, θα πρέπει να πω, με το ακανθοδέστερο ίσως πρόβλημα για την ΚΑΠ μετά το 2013. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μιλούν για μια ε, ενιαία πρημοδότηση αναεπιφάνεια από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως θα έχει τεράστια ε, μετατόπιση πόρων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως συνέπεια. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, έχουμε εδώ την υποστήριξη και τη συνεργασία όλων των κρατών μελών και ίσως ε, θα μπορούσαν οι πληρωμές να προσαρμοστούν, ε, να διαμορφωθούν με βάση αντικειμενικά κριτήρια τα οποία θα με τις διαφορετικές συνθήκες, αλλά ταυτόχρονα θα καλύπτουν και τις διαφορές σε σχέση με το, με την, με το κόστος παραγωγής. Κυρίε και κύριοι, συχνά μιλούμε για το κόστο στην παραγωγή, το κόστο τη γεωργία, το κόστο των τροφίμων. Όμω δεν πρέπει να λησμονούμε και το, ε, την προσθέμενη αξία, το τι προσφέρει η γεωργία για την Ευρώπη, για τον Ευρωπαίο. Το ότι μπορούμε να έχουμε δηλαδή τα καλύτερα, τα φθηνότερα, τα πιο θρεπτικά και τα πιο υγιεινά τρόφιμα, όχι μόνο στον κόσμο, αλλά σε ολόκληρη την ιστορία του ανθρώπου. Και ταυτόχρονα μια υγιή γεωργία, ε, μια ύπεθρο ε, με την πολυμορφία της, με την ποικιλία της και έναν γεωργό σε απασχόληση όπως το προτιμάει, όπως θέλει μας στην Ευρώπη. Έτσι μπορούμε να έχουμε την καλύτερη, πιστεύω, ε, σχέση κόστους και αποτελέσματος, τα καλύτερα ωφέλη από την κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε λοιπόν πάντα δίνοντα το λόγο στου γεωργού και εκπρόσωπους ε, της Υπέθρου. Ραφαέλ Ερνάντες, λοιπόν, θα είναι ο επόμενος ομιλητής μας, μέλος ε, ε, του Ευρωπαϊκού Συντονισμού ε, Βία Καμπεσίνα. Έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να μιλήσουμε εξ ονόματος ε, ε της ε, Βίακαν Πεσίνα και ε, εξ ονόματος του Μάρτιν Χάουσλινγκ. Είναι ε, μια ευκαιρία αυτή που μας δίνεται και θέλουμε να την αξιοποιήσουμε πρώτα απ' όλα για να για να μιλήσουμε για την οργάνωση αυτή ε, γεωργών από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία που έχει το γεγονό ότι μα δίνει αυτή την ευκαιρία για να μεταφέρουμε τι τις προτάσεις μα, γιατί πραγματικά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια στιγμή μεταβατική και θέλουμε να λάβουμε τι ευθύνε μα και ταυτόχρονα θα θέλαμε επίσης με την προσοχή στις δικές σας ευθύνες, ε, αλλά και στη δέσμευση των μελών της Επιτροπής Γεωργίας που θέλετε να συμβάλλετε ε, προς τη βελτίωση των συνθήκων διαβίωσης ε, των γεωργών ανδρών και γυναικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στο τέλος μιας φάσης της κοινή αγροτικής πολιτικής που απέτυχε όσον αφορά ορισμένες πτυχές. Και όπως σαφώς αυτοί που πλήττονται είναι οι γεωργοί και οι καταναλωτές. Είναι λοιπόν σημαντικό να το τονίσουμε το στοιχείο αυτό, διότι ορισμένοι από τους στόχου που έχουν τεθεί δεν έχουν επιτευχθεί. Όπως ε, για παράδειγμα η εγγύηση ενός ισότιμου ε, επίπεδου διαβίωσης σε αυτούς που ζουν στην Ήπεθρο, σταθεροποίηση των αγορών, εγγύηση προς τον καταναλωτή την πρόσβαση στα αγαθά και βλέπουμε το πώς ε, ο κόσμος τη υπαίθρου, ο αγροτικό πληθυσμό γυράσκει, όλο και περισσότερο, ε, ε, με όλο και περισσότερη δυσκολία εντάσσονται στο επάγγελμα οι νέοι, με αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, εμείς θέτουμε την εξή πρόταση, η οποία σχετίζεται και ε, αφορά το εξή. Πέραν τη ασφάλεια ε, του εφοδιασμού τροφίμων, κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και μιλάμε για ε, επισητιστική διατροφική κυριαρχία. Θα θέλαμε λοιπόν από το 2013 και εξή να μην χρησιμοποιείται ο όρος ΚΑΠ, αλλά να μιλάμε για, τη για την κοινή γεωργική και επιστηστική και πολιτική στο τομέα των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση λοιπόν αυτή έχει να κάνει με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και με βάση και την ατζέντα 2020 ε, που αναφέρατε, ε, την αλλαγή του κλίματος. Το καθορισμό λοιπόν ενός ε, οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού μοντέλου που να είναι αηφόρο. Ο κόσμος της γεωργίας λοιπόν προσφέρει απασχόληση στα άτομα που δεν έχουν. Το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει να δούμε είναι το εξή. Για ποιον γίνεται η παραγωγή, πώς γίνεται η παραγωγή και ποιος παράγει. Είναι σαφές ότι ο στόχος Τη παραγωγή, ε, η απάντηση στο ερώτημα γιατί γίνεται η παραγωγή, στόχος είναι ε, η ε, κάλυψη των αναγκών διατροφής του πληθυσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και όχι απαραίτητα η εξαγωγή. Γιατί αν προσανατολίζουμε την παραγωγή προς τι εξαγωγέ, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τι θα γίνει. Δεν θα, θα είναι αβάσταχτη πλέον η κατάσταση, διότι ε, ε, ε, ε έχουμε την εξάρτηση ε, από τα καύσιμα για, το, για, για, για, τις μεταφορές, για παράδειγμα, και θα είναι αβάσταχτη η κατάσταση. Δεύτερον, πώς θα γίνεται η παραγωγή. Ποιος θα είναι ο παραγωγός. Είναι σαφές ότι η, η οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να απαντήσει στην πρόκληση αυτή. Εφόσον η διατροφή είναι και πολιτική πρόκληση και τεχνολογική πρόκληση και πρόβλημα διανομής αλλά και ε, πρόβλημα που έχει να κάνει με την αύξηση, ε, με την ανεξέλεγκτη αύξηση παραγωγικότητας. Και ακριβώς εδώ ε, απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που ασκούν την πολιτική εξουσία και έχουν την ευθύνη να δώσουν απαντήσεις στις ανησυχίες μας αυτές. Και τρίτη απάντηση που θα πρέπει να δοθεί είναι το πώ θα γίνει η παραγωγή. Εμεί από την πλευρά τη δική μα οργάνωση πιστεύουμε ότι προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση ε, του αντίκτυπου ε, στην ε, αλλαγή του περιβάλλοντος, στην διασφάλιση της βιοπικιλότητας, στην, διατήρηση του, στην αντικατάσταση του υφιστάμενου μοντέλου, στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος. Και εδώ έχουμε ορισμένα στοιχεία κλειδιά. Πρώτον, σταθερέ τιμέ και ανταποδοτικέ που να επιτρέπουν στο Γεωργό να μπορεί να ζει από την ε, δραστηριότητά του τη γεωργική. Επίση, και το αναγνώρισε και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρόσφατα αναφέρθηκε σε μια ανακοίνωση για μια καλύτερη αλυσίδα τροφίμων και εφοδιασμού στην Ευρώπη. Αναγνωρίστηκε λοιπόν η, η, η κατάχρηση από τις μεγάλες αλυσίδες διανομής, η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Γι' αυτό εδώ θέτουμε συγκεκριμένες προτάσει. Πρώτα απ' όλα, τα νέα πλαίσια θα πρέπει να ε, συμπεριλαμβάνουν μέτρα ρύθμιση της παραγωγής και ρύθμιση των γεωργικών αγωγών. Αυτό είναι βασικό κατά την άποψή μου. Επαναπροσανατολισμός λοιπόν αυτών των παραγωγών που είναι πλεονασματικές και αύξηση των ε, ελληματικών παραγωγών. Θα πρέπει να ε, καταργηθεί η έλλειψη διαφάνειας σε όλο το μήκος της ε, αλυσίδας τροφίμων, ε, να υπάρξει ε, καλύτερος επιμερισμός των εσόδων, καθόλου το μήκος της αλυσίδας. Άρα γι' αυτό θα πρέπει να θεσπιστούν ελάχιστες τιμές των προϊόντων τη στιγμή της κρίσης. Γι' αυτό απαιτείται ο περιορισμός ή η αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος ανταγωνισμού. Θα πρέπει να περιοριστούν ε, τα κέρδη καθ' όλη το μήκο τη αλυσίδα. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε αυτή την άνηση κατάσταση. Και αυτό θα πρέπει, θα πρέπει λοιπόν να γίνει νέε διαπραγματεύσει με βάση τις αρχές του fair play. Ε, της ισοτιμίας και της δικαιοσύνης. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε ε, και να δώσουμε κίνητρα για ε, άμεση εμπορία. Αυτό όμως θα απαιτήσει ένα κανονιστικό πλαίσιο όπου να δίδεται περισσότερος πρωταγωνιστικός ρόλος στο γεωργό και στον καταναλωτή. Το δικαίωμα του καταναλωτή είναι να μπορεί να επιλέγει τα τρόφιμα τα οποία θα καταναλώσει και το από ποια παραγωγή προέρχονται. Και επίσης να ξέρουμε και το ίχνος του άνθρακα του συγκεκριμένου προϊόντος. Καταλαβαίνετε, 8.000 ε, ε, χιλιόμετρα κατά μέσο όρο διανύουν τα τρόφιμα μέχρι να φτάσουν στα ράφια των μεγάλων σούπερ, μάρκετ. Όσον αφορά το εξωτερικό επίπεδο, και εδώ μιλάμε για την οργάνωση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε σχέση πάντα με την, με την αγροτική πολιτική. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι Ακριβώς η κυριαρχία ε, στον τομέα της διατροφής δεν σημαίνει αυτάρκεια, ούτε κλείσιμο των συνόρων, ούτε ε, με τοπική αντιπαράθεση απέναντι σε οποιαδήποτε ε, παγκόσμια συναλλαγή. Κάθε περιοχή του κόσμου έχει το δικαίωμα να παράγει τα δικά της προϊόντα και να μπορεί να τα θέτει σε εμπορία. Όμως, εμείς στην οργάνωσή μας πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό ότι είναι πολύ σημαντικό θέμα ε, η διατροφή και δεν μπορεί να εξαρτάται από τις αγωγές. Σε κάθε περιοχή του κόσμου ε, η βασική, τα βασικά είδη διατροφής θα πρέπει να παράγονται ώστε το τον περισσότερο σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό κάθε περιοχή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να προστατεύει τον εαυτό της από τις εισαγωγές ε, χαμηλού κόστους που καταστρέφουν την τοπική παραγωγή. Με βάση αυτά διεκδικούμε τη θέσπιση ε, επιπέδων ε, παραγωγής ε, για τους δασμούς που να έχει σχέση και με το επίπεδο της ευρωπαϊκής παραγωγής. Και δεν θέλω να πω για παράδειγμα, πρόσφατα υπεγράφει συμφωνία σύνδεσης με το Μαρόκο. Και εκεί όχι μόνο δεν συμβάλλει αυτή η συμφωνία στο να καταναλώνουν πιο φτηνά τα οποροκυπευτικά οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά θα επιδεινώσει τα πράγματα. Και κάτι άλλο, άλλο παράδειγμα σας δώσω η μείωση των δασμών στην, περίπτωση των... της μπανάνας, για παράδειγμα. Δεν θα ωφελήσει ούτε του Ευρωπαίου καταναλωτέ, ούτε του παραγωγού στη χώρα προέλευση. Ε, ένα κυβότιο μπανάνε. Ε, όπου ε, πληρώνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 20 ευρώ. Στην Κεντρική Αμερική οι παραγωγοί παίρνουν ε, μόλις 3 δολάρια και καταλαβαίνετε κάθε φορά ε, εκεί η κοινωνική κατάσταση επιδεινώνεται. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας. Και εσείς ε, ε κυρίες και κύριοι μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να ακολουθείτε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ε, έχουμε μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια ευκαιρία για να διορθώσουμε τα πράγματα. Τα κριτήρια τα οποία ακολουθούνται για, την παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ακολουθούνται και να ισχύουν και για τι χώρε από τι οποίε ε, αγοράζουμε τα προϊόντα του. Για να βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο, οι συνθήκε παραγωγή. Και αυτό δεν είναι καλό μόνο για μα, αλλά και για αυτέ τι χώρε. Γι' αυτό σα λέω ότι είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίσουμε το εξή ότι αυτά τα μέτρα δεν ωφελούν ούτε εκείνου ούτε εμά. Πέντε μεγάλε πολυεθνικέ ωφελούν στην περίπτωση τη μπανάνα, που ελέγχουν το 95% ε, του παγκόσμιου εμπορίου μπανάνα. Ε, γι' αυτό δεν χρειάζονται να, να ληφθούν μέτρα προ την κατεύθυνση αυτή. Ε, για αυτέ δηλαδή. Και τέλο να σα πω ότι θα πρέπει να δούμε τι άμεσε ενισχύσει που παίρνουν οι παραγωγοί. Εμεί η παραγωγή παίρνουμε από την αγορά μόλι το 20% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 20% ε, αυτού που πληρώνουν οι καταναλωτέ. Με διαφορέ 400, 500 και 1000%. Λοιπόν, ανάμεσα σε εκείνη τη, ανάμεσα απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, για να διατηρήσουμε τι δραστηριότητέ μα στην ε, Ήπεθρο, χρειαζόμαστε ενίσχυση. Γι' αυτό θα πρέπει να προσανατολίσετε αυτέ τι ενισχύσει στι εκμεταλλεύσει που ε, έχουν αποδείξει ότι παίζουν το ρόλο του σε κοινωνικό επίπεδο, σε περιβαλλοντικό επίπεδο, δημιουργούν θέσει απασχόληση, κρατούν τον κόσμο στην Ήπεθρο και στι γεωργικέ δραστηριότητε. Και τέλο να σα πω ότι αυτό το μοντέλο το οποίο προτείνεται, σχετίζεται, προτείνουμε, σχετίζεται όχι μόνο με τα συμφέροντα των γεωργών, αλλά και με ε, τα, διάφορα, τις τα διάφορα φάσματα τη κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρόσφατα υπεγράφει μία δήλωση για, την, ε, για το τρόφιμα που αποτελεί ε, σαφέ παράδειγμα όχι μόνο αυτού που ζητούν οι Γεωργοί, αλλά αυτό που ζητάει η κοινωνία των πολιτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σα ευχαριστώ ε, που με ακούσατε. Ευχαριστούμε τον Ραφαέλ Ερνάντες και δίνω τώρα το λόγο στον Πίτερ Κένταλ πρόεδρο της National Farmer Union, ο κύριος Κέντελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς την Επιτροπή. Με προσκάλεσε εκ μέρους της Εθνικής Ένωσης της Αγγλίας Ουαλίας να σας μιλήσω, αλλά επίσης και για το γεγονό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο προ τη συζήτηση για το μέλλον τη κοινωνική πολιτική. Εγώ προσωπικώ είμαι γεωργό 20 μίλια δυτικός του Κέμπριτζ και βορείος του Λονδίνου περίπου. Είμαι γεωργός που πιστεύω πως θα με διαδεχθούν τα παιδιά μου κάποια στιγμή και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά και σε επόμενες γενναίες. Κάνουμε λοιπόν ε, τη δουλειά μας ε, όσο καλύτερα μπορούμε και επενδύουμε για το μέλλον. Ε, εάν κοιτάξουμε λοιπόν τις μεγάλες προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι σημαντικό ασφαλώ, ο γεωργό να έχει και την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση, να μπορεί να προγραμματίσει για το μέλλον και να προβαίνει σε μακροχρόνιες επενδύσεις. Αυτό πιστεύω σημαίνει ταυτόχρονα και χρήση των επενδύσεών μας. Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να περάσουμε από την οικονομία του ίδρογον άνθρακα στην οικονομία, στην οικονομία του υδατάνθρακα περισσότερο. Δηλαδή να είμαστε σε θέση να παράγουμε τρόφιμα τα οποία θα μπορούν να θρέψουν ολόκληρο τον κόσμο. Η γεωργία είναι, πιστεύουμε, κεντρικός παράγων σε αυτή αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών που εντόπισε νωρίτερα και ο συνάδελφο κ. Λάιον. Ο Γεωργό, ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, πιστεύω, και έχουμε εδώ και από το Άλστερ, από τη Βορεια Ιρλανδία δηλαδή, γεωργού από ό,τι γνωρίζω, δεν θα πρέπει να εξαρτάται από την υποστήριξη κάποιου προϋπολογισμού. Θέλουμε δηλαδή η αγορά να είναι πιο δίκαιη απέναντι στο γεωργό και να τον μεταχειρίζεται ισότιμα. Εάν κοιτάξουμε την ευρωπαϊκή οικονομία γενικότερα, φαίνεται ότι ο φορολογούμενος καλείται να στηρίξει την παραγωγή μας. Τι γεωργικέ μα αγορέ. Πρέπει να βρούμε καλύτερο τρόπο λειτουργία λοιπόν αυτών των γεωργικών αγορών, γιατί ο γεωργό δεν θέλει να εξαρτάται από την στήριξη του φορολογούμενου. Δεν θέλει να εξαρτάται πλην όμω, πλην όμω, ακούσατε να γίνεται λόγο ήδη για την κρίση σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται η στήριξη, χρειάζεται ο παραγωγό να υπάρχει τώρα, να τον στηρίξουμε τώρα και θα χρειάζεται να διατηρηθεί να διαφυλαχθεί η λειτουργία του και για το μέλλον. Η ΚΑΠ αυτό το ρόλο καλείται να επιτελέσει. Έχει εξασφαλίσει σημαντική πρόοδο, έχει επιτρέψει στις αγορές μας να προχωρήσουν και είναι, πιστεύω, θετικό ότι έχουμε, ότι έχουμε δεσμευθεί να ε, καταργήσουμε τις επιστροφές της εξαγωγές. Είμαστε μια πλούσια ένωση, ένα πλούσιο σύνολο χωρών Έχουμε πλεονασματικά προϊόντα τα οποία μπορούμε να τα διαθέσουμε σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές, αλλά όχι με ε, επιδότηση των ε, εξαγωγών μας, γιατί αυτό είναι και εσφαλμένο οικονομικά, αλλά και ανήθικο. Πρέπει να βρούμε διαφορετικό τρόπο να απορροφήσουμε αυτή την επιπλέον παραγωγή. Έτσι λοιπόν, κοιτώντα τη σημασία της γεωργίας και την σημασία της διαφύλαξης της για το μέλλον, πρέπει ασφαλώς να βρούμε τον τρόπο να εξασφαλίσουμε τη συνέχιση της χωρίς όμως τραύλους των αγορών. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συζητήσει τον τρόπο ακριβώς με τον οποίο μπορεί να διαφυλαχθεί ε, ο γεωργός χωρίς την υποστήριξη του πρώτου πυλώνα, χωρίς την ρητή υποστήριξη του πρώτου πυλώνα, χωρίς τον, προσα... τον προστατευτισμό τον οποίο έχουμε γνωρίσει τελευταία χρόνια, γιατί μας θυμίζει σε όλους βέβαια αυτός ο προστατευτισμός ότι υπάρχουν χώρες σε όλο τον κόσμο που έχουν καταφύγει σε πιο προστατευτικές πολιτικές ε, αλλά έκαναν λάθος με τον τρόπο αυτό και γι' αυτό πιστεύουμε ότι χωρίς να εγκαταλείψουμε την γεωργία εκτεθειμένη 100% στις συνθήκες της αγοράς, θα πρέπει να είμαστε σε θέση ως Ευρωπαϊκή Ένωση να εξηγούμε στον καταναλωτή μας, στον φορολογούμενο δηλαδή, γιατί χρειαζόμαστε μια γεωργική πολιτική πιο ισχυρή και κοινή μέσα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν είναι, έχει ως όρο απαρέκλειτο τη διατήρηση των ε, άμεσων πληρωμών στον πυλώνα όσο μπορούν οι ανταγωνιστές από όλο τον κόσμο να έχουν τη ε, δυνατότητα πρόσβαση στην αγορά μας και να πιέζουν τόσο πολύ τα εισοδήματα των παραγωγών μας. Για όλο αυτό το διάστημα, μέχρι τότε δηλαδή που θα σταματήσει αυτή η πίεση, θα πρέπει να διατηρηθούν οι άμεσες πληρωμές. Όταν σταματήσουν ε, οι πιέσεις από, τις αμερικανικές, από την αμερικανική παραγωγή, όταν σταματήσει η πίεση που λέει να, πει, να παράγεις λιγότερο, λιγότερα τρόφιμα γιατί αλλού είναι πιο φτηνά, χρειαζόμαστε ακόμη αυτές τις πληρωμές από τον πρώτο πυλώνα. Διαφορετικά θα περάσουμε 7 χρόνια ε, ισχνών αγελάδων, όπως θα περάσουμε και 7 χρόνια παχαίων αγελάδων, αλλά θα πρέπει να είμαστε σε θέση να εξισώσουμε τις συνθήκες της πρώτης με τη δεύτερη εφταετία. Πρέπει λοιπόν, χάρη στην ΚΑΠ, να είμαστε σε θέση και τα χρόνια των παχαιών αγελάδων να τα ε, αξιοποιήσουμε κατά τρόπον μακροπρόθεσμο, δηλαδή φυτεύοντας λιγότερο στις, ε, στα χωράφια μας και δουλεύοντας με προγραμματισμένο τρόπο έτσι ώστε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στην περίοδο της, ε, των πλεονασμάτων σε μια σταδιακή απεξάρτηση από τις πληρωμές του πρώτου πυλώνα. Εγώ θα ήθελα να φτάσει η στιγμή που θα μπορούμε να δούμε αγορές που θα λειτουργούν ελεύθερα και όπου θα μπορεί μέσα σε αυτές ο Γεωργός να προσφέρει την υπηρεσία του. Είναι απαραίτητο να ε, εξισορροπηθούν οι αυξήσει των τιμών, όπω είπα, όθηκε νωρίτερα, έχουμε αύξηση τιμών στον ε, καταναλωτή 47%, ενώ ήταν μόνο 27% για τον παραγωγό. Αυτό δείχνει ότι οι αγορέ έχουν ξεφύγει από το μέτρο και αν θέλουμε να έχει ο παραγωγό ένα κομμάτι ε, δίκαιο από αυτές τις αγορές, θα πρέπει αυτές οι αγορές να λειτουργήσουν οι ίδιες κατά τρόπο δίκαιο και ισότιμο και πιστεύω ότι εδώ μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ε, δική της συμβολή Όπω ε, παραδείγματι με ένα παράδειγμα που συστήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ε, δυνατότητα εξασφάλισης δίκαιων τιμών, ιδιαίτερα για το γαλακτοκομικό τομέα, γιατί ιδιαίτερα στην Βρετανία ξέρουμε ότι ο τομέας ο γαλακτοκομικός έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για την σύντησή μας, για, για την παροχή ενό βασικού αγαθού, ενό βασικού τροφίμου, αλλά και για τη φύλεξη του ίδιου του τοπίου του Βρετανικού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε μάκρο, μακροπρόθεσμα σταθερέ τιμέ για τον παραγωγό, ώστε να μην... Ε, ε, ροκανίσετε διαρκώς το περιθώριο κέρδους από τον ε, Λιάνο Πολιτή, από το σούπερ μάρκετ δηλαδή. Και ταυτόχρονα θέλουμε να έχουμε και σήμανση σαφή, να μπορεί ο καταναλωτής να διαγιγνώσει ότι είναι υψηλέ οι προδιαγραφές ποιότητας στο ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γεωργική παραγωγή εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην έχουμε αυτό το συνονθήλευμα πληροφοριών ή μάλλον καλύτερα ένα μείγμα ε, προϊόντων η διάθεση του καταναλωτή που όμως δεν του επιτρέπει να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να περάσουμε πάλι στη συζήτηση για τη χρηματοδότηση κοινή γεωργικής πολιτικής και τη σημασία της ύπαρξης της κοινή γεωργικής πολιτικής. Το κρίσιμο στοιχείο για την επιβίωση της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι η κοινή χρηματοδότησή της. Η συγχρηματοδότηση θα σήμαινε οψοδρόμηση. Ανησυχώ ιδιαίτερω διότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, εάν δηλαδή ε, κληθούν τα κράτη-μέλη μεμονωμένα να συμπληρώσουν την, ε, τις πληρωμές για τη γεωργία τους, αυτό πολύ γρήγορα θα φέρει και το τέλος της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Όχι της κοινής γεωργίας, της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει μόνη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, αντιδράσει σε αυτό. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μεγάλες προκλήσεις και θα έχουμε τα επόμενα 20, 30, 40 χρόνια ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση, όπως είπε και ο κύριος Λάιο νωρίτερα, ότι με δεδομένες τις κλιματικές αλλαγές, δηλαδή με επιδείνωση των φυσικών συνθήκων, θα έχουμε μεγαλύτερο πληθυσμό ακόμη να, να θρέψουμε στα επόμενα 30, 40 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να σας μιλήσω. Bene, grazie. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Πίτερ Κέντεν. Τελειώνουμε λοιπόν αυτό τον πρώτο γύρο ε, με τους εμπειρογνώμονες ε, του κόσμου της Γεωργίας και να δώσω το λόγο στον Άλμπερτ Γιάν Μάτ, ε, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ στις Βρυξέλλες. Άλμπερτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, με, μεγάλη ευχαρίστηση, ξαναβλέπω παλιούς συναδέλφους και χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον της ΚΑΠ. Θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη της Επιτροπής σας για την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας διότι έτσι αναλαμβάνεται ένα σημαντικότατο ρόλο συνομοθέτη στα πλαίσια της κοινή γεωργικής πολιτικής. Εγώ μιλώ εξ ονόματος ε, ε, πολλών ε, γεωργών και περιβολάριδων της Ολλανδίας που θεωρούν ότι είστε οι καλύτεροι εγγυητές για την ΚΑΠ και σας ευχαριστούν γι' αυτό. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη νέα στρατηγική ΚΑΠ 2020. Εσείς διαμαρτυρηθήκατε πολύ έντονα λέγοντας ότι δεν μιλάμε καθόλου για γεωργία, δεν μιλάμε καθόλου για τα πορικυπευτικά, δεν μιλάμε καθόλου για γεωργία. Και ας επανέλθουμε στην ΚΑΠ. Η ΚΑΠ είναι απολύτως απαραίτητη για το γεωργικό ευρωπαϊκό τοπίο. Εμείς γνωρίζουμε ότι ο αγροτικός πληθυσμός αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Αυτοί οι αγρότες όμως είναι υπεύθυνοι για τη γεωργική παραγωγή, οπότε είναι απαραίτητο να τους διατηρήσουμε, να διατηρήσουμε το τοπίο, για το οποίο παίζουν σημαντικότατο ρόλο οι αγρότες, οι οποίοι παράγουν μέσα από τις καλύτερες συνθήκες στον κόσμο, διότι πρέπει να περιφρουρήσουν τόσο το, και να διαφυλάξουν τόσο το περιβάλλον όσο και την βιοπικιλότητα. Σε πολλά κράτη-μέλη όμως η, κατα... η πίεση είναι τεράστια πάνω στους γεωργούς ε, και της χώρας μου συμπεριλαμβανομένης και ακούμε ένα σωρό κριτικές για τον προπολογισμό και για τα κονδύλια. Η ΚΑΠΑ όμως έχει απόλυτη ανάγκη αυτού του ευρωπαϊκού προπολογισμού και είναι ουσιαστικότατο μετά το 2013 να έχουμε έναν επαρκή γεωργικό προϋπολογισμό. Συμφωνώ απόλυτα με όσα μας είπε ο αντιπρόεδρος, ο, προ, της ΚΟΠΑ και ό,τι μας είπε και ο Πίτερ Κέντελ. Για την Ολλανδική οργάνωση, εγώ θα ήθελα να αναφέρω μερικά σημεία, τα οποία είναι ουσιαστικότατα για μας. Εμείς θεωρούμε ότι η μεταρρυθμισμένη ΚΑΠΑ θα έπρεπε να προβλέπει την ανταμοιβή των γεωργών για ό,τι κάνουν και για την βιοποικιλότητα και για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Κάτι το οποίο και πραγματικά τους πολίτες αλλά για, τους, για, για τη διατήρηση των οποίων και τη συντήρησή τους δεν αμείβεται κανείς. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την ΚΑΠ προς αυτήν την κατεύθυνση και στον πρώτο πυλώνα. Αυτό θα πρέπει να γίνει μέχρι το 2013. Χρειάζεται επίσης να είμαστε ιδιοκτήτες των γεών μας. Θα πρέπει να αποφύγουμε να συνεχίζουμε να κατακαιρματίζουμε το γεωργικό τοπίο όπως γίνεται σήμερα, διότι αυτό θα έχει άσχημες συνέπειες και για την γεωργική παραγωγή, αλλά και για το τοπίο και για τη βιοπικιλότητα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να προσέξουμε ούτως ώστε όλες οι πράσινες υπηρεσίες να συνεχίζουν να παρέχονται αλλά και να ανταμείβονται. Η γεωργική παραγωγή λοιπόν και τροφιμική ασφάλεια. Αυτό θα πρέπει να γίνεται στα πλαίσια, σε μια αγορά ε, που βρίσκεται εν πλήρη εξελίξη. Γκρεμίζονται οι δασμοί και τα εμπόδια, αλλά θα γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε εμείς ε, ικανοί να ανταγωνιζόμαστε με τα προϊόντα μας στις παγκόσμιες αγορές και χρειαζόμαστε γι' αυτό ενισχύσεις. Γνωρίζουμε ότι μέχρι το 2050 θα, έχουμε, θα πρέπει να έχουμε μία αύξηση 70% της παραγωγής. Και στο αεροβαρόμετρο διαπιστώσαμε ότι οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η ΚΑΠ θα πρέπει να, να, εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο. Κανένας λοιπόν δεν αμφισβητεί ούτε την ΚΑΠ ούτε τον προπολογισμό της. ο κόσμος ε, τα βλέπει όλα αυτά με πολύ καλό μάτι. Θα πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε και την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Είναι σημαντικότατα αυτά για την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων στο μέλλον. Αν εμείς έχουμε όλο ένα λιγότερες ε, πρώτες ύλες και μας ζητούν όλο ένα περισσότερο γεωργικά προϊόντα, θα πρέπει να μπορέσουμε να απαντήσουμε με καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να παράγουμε περισσότερο, με λιγότερα μέσα και με αηφορία. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε πρωτοπορία στον κόσμο, αυτό τουλάχιστον εμείς θέλουμε στην Ολλανδία, διότι εμείς ε, είμαστε οι δεύτεροι ε, σε μέγεθος ε, παραγωγή τροφίμων. Γι' αυτό λοιπόν ε, κοιτάξαμε να κάνουμε ό,τι μπορούσαμε από συμφωνίες και συμβάσεις για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε 2% μείων ενέργεια να καταλώνουμε, 30% μείωση εκπομπών αερίων μέχρι το 2015 και 20% να είναι το ποσοστό της αηφόρου φόρου ενέργειας που χρησιμοποιείται στη Γεωργία. Αλλά κύριε Πρόεδρε υπάρχουν ένα σωρό τομείς όπου η γεωργική παραγωγή δεν είναι το optimum και για να συνεχίσουμε να, να προστατεύουμε το τοπίο χρειάζεται να λάβουμε παραπάνω μέτρα και να δώσουμε τα απαραίτητα κονδύλια. Μιλάτε εσείς για διαχείριση των αγορών. Για πολλές γεωργικές παραγωγές για το τοπίο και για γεωργικές παραγωγές μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή βοηδή, γάλα, ζαχαρότευκλα, πατάτες και αμυλώδη. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ένα σχέδιο για ένα νέο μέσο, μέσο ε, Οργάνωση των αγορών, ε, για τα δημητριακά επίσης, ούτως ώστε να έχουμε σταθερές τιμές και τη σωστή πλαισίωση. Και όταν υπάρχει η υπερπαραγωγή, το, τα προϊόντα, τα, τα πλεονάσματα να μπορούν να διοχετεύονται στην αγορά των βιοκαυσίμων. Και ελπίζουμε σε αυτό να μας βοηθήσει και το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, παραγωγή τώρα. Η παραγωγή και οι σχέσεις τους με τα σούπερ μάρκετ. Με τα μεγάλα δίκτυα διανομής δηλαδή. Θα πρέπει να καταφέρουμε να συνεργαστούμε καλύτερα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η παραγωγή θα πρέπει να οργανωθούν σε, σε κλαδικές οργανώσεις παραγωγή τροφίμων για να αντιμετωπίσουν την μεγάλη διανομή. Υπάρχει η δεσπόζουσα θέση των σούπερ μάρκετ, είναι απαράδεκτη κατάσταση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ομαδοποίηση της προσφοράς, την ομαδοποίηση των γεωργών και να μας βοηθήσει η Κομισιόν γι' αυτό. Θα πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι χωρίς τους Ευρωπαίους παραγωγούς η προσφορά και η διαφορετικότητα θα εκλείψουν. Χρειάζεται λοιπόν οι κανόνες του ανταγωνισμού να προσαρμοστούν ώστε αν ο παραγωγός συνάπτει συμφωνίες με τα σούπερ μάρκετ αυτή η συμφωνία να είναι πιο διαρκής και να υπάρχει μια σωστή κατανομή των δαπανών σε όλη την αλυσίδα της διανομής. Για τις γεωργικές επιχειρήσεις θα πρέπει εμείς να διασφαλίσουμε ότι η αγροτική πολιτική θα παραμείνει κοινή. Θα, δεν θα πρέπει να οδηγήσουμε στην επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ. Τότε οι Γεωργοί, οι Ευρωπαίοι αγρότες θα είναι ανταγωνιστές μεταξύ τους και δεν θα μπορούν να παράγουν για την Ευρώπη και για τον υπόλοιπο κόσμο. Χρειάζεται λοιπόν κοινή αγροτική πολιτική με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τα υψηλά στάνταρ και για τις ε, και για το περιβάλλον ε, και για την ποιότητα των προϊόντων. Είναι και θέμα κουλτούρας. Πρέπει λοιπόν να παραμείνει κοινή αγροτική πολιτική με τη βοήθειά σας. Ευχαριστώ Άλμπερτ. Μπορείς να μετράς ε, με τη βοήθειά μας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε. Τελείωσε λοιπόν το πρώτο κομμάτι των τοποθετήσεων και ξεκινάει η συζήτηση. Ένα, μια πρώτη συζήτηση να δώσω το λόγο πρώτα στους συντονιστές των ομάδων και μετά σε όλους όσους ε, ζήτησαν να μιλήσουν. Μετά από αυτήν την ε, σύντομη συζήτηση θα έχουμε ένα δεύτερο πάνελ τοποθετήσεων και μετά θα έχουμε το κλείσιμο της συζήτησης. Ξεκινάω λοιπόν από τους σοσιαλιστές, τον Λουίς Κάπουλας Σάντος. Έχεις το λόγο Λουίς. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας ε, τον εισηγητή μας ε, για την, ε, για την παρουσίασή του. Πραγματικά μας παρουσίασε συγκεκριμένες παρατηρήσεις και είναι πάρα πολύ χρήσιμο το έγγραφο εργασίας. Καταβλήθηκε λοιπόν μεγάλη προσπάθεια και γι' αυτό ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους μας και ιδιαίτερα ε, τα πρώην μέλη του Κοινοβουλίου. Με μεγάλη χαρά ε, υποδεχόμαστε κάθε φορά πρώην συναδέλφους. Κυρίε και κύριοι, όλοι γνωρίζουμε ότι η στιγμή που διανύουμε είναι δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη και όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο η οικονομία και η κοινωνία αυτή τη στιγμή διανύουν δύσκολες στιγμές. Και ακριβώς επειδή οι στιγμές είναι δύσκολες, ε, ταυτόχρονα δημιουργούνται κάποιες ευκαιρίες. Και εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να προβούμε στη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής που είναι ε, μία από τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βέβαια στέφει από μεγάλη επιτυχία, αλλά που πρέπει να την προσαρμόσουμε στη σημερινή πραγματικότητα. Πραγματικότητα που είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ε, μια, μια πραγματικότητα όπου σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γίνονται ε, δημοσιονομικές περικοπές, δεν προβλέπονται αυξήσεις των προπολογισμών, ενώ αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός των δικαιούχων, αυτών που αποφελούνται από τις ενισχύσεις της ΚΑΠ, η οποία με τον τρόπο αυτό διαθέτει όλο και λιγότερα κονδύλια. Γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Πάντως είμαι σίγουρος για το ότι τα ευρωπαϊκά όργανα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την τεράστια πρόκληση. Κοίταξε κύριε Πρόεδρε, εγώ είμαι αισιόδοξο από τη φύση μου. Και, και, αλλά και σε αυτή τη στιγμή είμαι αισιόδοξο. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι όλοι ε, έχουμε κάποιες ε, κοινέ απόψεις, ένα κοινό παρονομαστή. Είναι σίγουρο ότι, είναι προφανές, ότι οι, οι, οι ομιλητές τόνισαν το ότι θα πρέπει πάντα να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική με την έννοια ότι πρέπει να απορρίψουμε κάθε προσπάθεια επανεθνικοποίηση. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει και να μην πέσουμε στην παγίδα τη πανεθνικοποίηση. Ε, Ζώντα τη σημερινή κατάσταση και τη σημερινή χρονική στιγμή, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν, δεν διαθέτουν απεριόριστου πόρους για να μπορούν να καλύψουν το δικό του μέρο στη συγχρηματοδότηση. Και ταυτόχρονα πρέπει να πούμε, να δούμε τι κοινή αγροτική πολιτική θέλουμε, πιο δίκαιη, πιο ισότιμη και περισσότερη νομιμότητα απέναντι στου πολίτε, στην κοινωνία των πολιτών. Αυτό τι σημαίνει. Αναδιάρθρωση τη αρχιτεκτονικής δομή τη ΚΑΠ. Και πρέπει να τολμήσουμε, να επιδείξουμε θάρρο. Γιατί κάθε φορά που γίνεται μια συζήτηση για το θέμα αυτό, τότε ακούμε φωνές υπέρ και κατά. Α, κοιτάξτε, εδώ ε, πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις ε, ε, διαφωνίες, γιατί δεν έχει νόημα να εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η διχοτόμηση. Η νομιμότητα των ενισχύσεων του πρώτου πυλώνα πρέπει να είναι η ίδια με, την, ε, με τις ενισχύσεις στα πλαίσια του περιβάλλοντος και του δεύτερου πυλώνα. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι δεν πρέπει να καταργήσουμε ούτε τον πρώτο ούτε τον δεύτερο πυλώνα, αλλά να διατηρήσουμε τι ενισχύσει με την ίδια νομιμότητα και στου δύο πυλώνε, έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη ζωή των ε, γεωργών και να μπορέσουμε να μειώσουμε το διοικητικό φόρτο εργασία τη στιγμή που δίδονται οι ενισχύσει αυτέ. Ο κύριο Λάιον ε, στο έγγραφο εργασία του αναφέρεται και ακολουθεί την οδό αυτή. Επίση, αισθάνομαι αισιοδοξία γιατί βλέπω ότι όλοι είναι υπέρ τη Ρύθμιση των αγορών. Όλοι συμφωνούμε στο ότι θα πρέπει να ρυθμίσουμε τι αγορέ. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι μέσα έχουμε στη διάθεσή μας και ε, τι, τι πακέτο θέλετε μέσων θα ε, χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις αγορές. Ταυτόχρονα πιστεύω στο ότι όλοι συμφωνούμε ε, ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη πέθρου και την οικονομική ε, αυτών των περιοχών με μέσα τα οποία ε, θα αφορούν για παράδειγμα την εγγύηση των εισοδημάτων. Όμως θα πρέπει να βελτιώσουμε και τις υποδομές, δηλαδή τις οδούς, τους δρόμους, ε, τις, ε, ε, τα συστήματα άρδευσης, ηλεκτροδότηση κτλ. Ζητώ λοιπόν τον κύριο Λάιον να, αναφέρει ότι θα πρέπει να καταργήσουμε το παλιό μοντέλο το οποίο δημιουργεί μόνο διαφωνίες. Θα πρέπει να επιδείξουμε την απαραίτητη τόλμη για να μπορέσουμε να καταργήσουμε αυτό το παροχημένο μοντέλο. Εμείς ως σοσιαλιστές συμφωνούμε με το ότι θα πρέπει όλοι να υποχωρήσουμε για να καταλήξουμε σε μια να τον ευρύτερη συμφωνία. Δεν μπορεί το Κοινοβούλιο να διαπραγματεύεται με το Συμβούλιο ε, για τα θέματα αυτά χωρίς να, μην μιλά, χωρίς να μιλά με μια ενιαία φωνή. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε με αυτή την ενιαία φωνή, γιατί μόνο με τον τρόπο αυτό θα είμαστε πιο ισχυροί στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Αυτό όμως με τη σειρά του απαιτεί να συμφωνήσουμε, να καταλήξουμε σε μια συνεργατική λύση. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σα πω συνοψίζοντα όλα αυτά με καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να σα πω ότι είμαστε στη διάθεση και των υπόλοιπων ομάδων για να ενισχύσουμε το έγγραφο αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ. Πολύ ωραίο αυτό το πνεύμα συνοχή και δίνω το λόγο ε, στον, ε, στον, στον Μισελ, εκπρόσωπο του ΕΛΚ. Έχει το λόγο, Μισελ. Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη καταρχάς εκ μέρους του Αλμπερτ ε, του στονιστού μας, γιατί δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ. Και εγώ προσωπικώς ε, στο συγγνώμη γιατί καθυστέρησα να έρθω στη συνεδρίαση, είχα ένα κατακτοπίσω ζήτημα. Είμαστε πεπισμένοι στην ομάδα μου ότι η κοινή γεωρική πολιτική που αποτελεί πλεονέκτημα ατού της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή οικοδόμηση. είναι θύμα σήμερα τη ε, επιτυχία τη πρέπει να το επαναλάβουμε, είναι όμω ταυτόχρονα ένα μέσον εξασφάλισης της ε, επιστηστικής αυτάρκεια τη Ευρώπη. Επιστηστικής αυτάρκεια μέσα σε συγκεκριμένα επίπεδα και προδιαγραφέ. Και το πρώτο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μα απασχολήσει και έναντι τη κοινή γνώμη, για να αιτιολογήσουμε την κοινή, την, το δημόσιο χρήμα που διαθέτουμε, τι δημόσιε ενισχύσει, είναι ότι προσπαθούμε να διαφυλάξουμε υψηλέ προδιαγραφέ, ευρωπαϊκές με κόστος κόστος, δηλαδή το επιπλέον κόστος στην παραγωγή, επιπλέον σε σχέση με το κόστος παραγωγής από τον υπόλοιπο κόσμο. Και επίσης θα ήθελα για το θέμα αυτό, το οποίο πιστεύω ότι είναι ουσιαστικά παραδεδεγμένο, δεν αμφισβητείται δηλαδή από κανέναν, είναι ότι η ευρωπαϊκή γεωργική παραγωγή είναι προσαρμοσμένη στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες και το περιβάλλον. Ταυτόχρονα λοιπόν θα πρέπει και να στηριχθεί οικονομικά όταν καλείται και να σέβεται περιβαλλοντικούς όρους που σημαίνουν ότι βρίσκεται σε σχέση δυσμενέστερο ανταγωνισμού, θα έλεγα σχεδόν αθέμητου, λέει ο μιλητής, σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και όταν στην Ευρώπη έχουμε μία παράδοση και παράδοση ζωής στην υπαίθρου και δρα ε, εργασία στην υπαίθρου, και έχει ένα ρόλο και διαφύλαξη της εδαφικής μας ε, χωροταξίας τη γεωργία. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες που πρέπει να προβάλλουμε ως λόγους για τη διατήρηση μιας ισχυρής κοινής πολιτικής. Φυσικά ε, θα πρέπει να παραδεχθούμε τις επικρίσεις, ότι διατυπώνονται επικρίσεις για τις μεγάλες, για τις ψηλότατες δαπάνες που έχουμε σε σχέση με τη γεωργία. Αυτό πάντα το βλέπουμε ούτως ή άλλως όταν υπάρχουν υψηλέ δαπάνες, το βλέπουμε και μέσα στα κράτη-μέλη, το βλέπουμε και σε σχέση με τις τοπικές περιφερειακές αρχές. Δεν θα πρέπει να ταραζόμαστε όταν ακούμε τέτοιου είδους κριτικές. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει είναι το ζήτημα της ρύθμισης των αγορών. Γιατί εδώ και μερικά χρόνια αναπτύσσεται μια θεωρία η οποία ε, τάση έχει την απορρίθμιση, απορρίθμιση η οποία και το 2007-2008 έδειξε ότι είναι ε, περιορισμένη με την ε, έξερση των τιμών στα γεωργικά και στα τρόφιμα και ιδιαίτερα με την κατάρρευση μετά των αγορών κάποιων γεωργικών προϊόντων και δι του γάλακτος. Άρα χρειαζόμαστε νέα μέσα, νέα εργαλεία και θα πρέπει να πείσουμε όλους τους γεωργούς, εγώ δεν λέω τους υπεύθυνους, τους ταγούς, γιατί αυτοί ίσως να το έχουν καταλάβει, αλλά τους γεωργούς, όλους τους γεωργούς της παλαιάς Ευρώπης, πρέπει να τους πείσουμε ότι όλα αυτά τα εργαλεία που είχαν σε θέση τα προηγούμενα χρόνια δεν μπορούν να ισχύουν στην Ευρώπη των 27. Γιατί έχει άλλη κλίμακα η Ευρώπη των 27. Δεν μπορεί να έχει την ίδια κλίμακα με την Ευρώπη των 6 ή των 12 ή των 15. Έτσι λοιπόν, άκουσα και άλλους που λέγανε ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα μέσα ρύθμιση των αγορών. Ερωτώ λοιπόν, ωραία, καμία καλή ιδέα έχετε να μας δώσετε για την λειτουργία αυτών των εργαλείων ή ποια εργαλεία για τη ρύθμιση των αγορών θα μπορούσατε να μας προτείνετε. Και ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Ευχαριστώ και τώρα δώσω το λόγο στον James Νίκολσον, εξ ε, των Ευρωπαίων Συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Um, Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι 17 Μαρτίου, είναι η ημέρα του ε, Αγίου Πατρίκιου στην Ιρλανδία. Εύχομαι λοιπόν σε όλες τις πατριώτες μου ε, χρόνια πολλά. Την ημέρα λοιπόν του Σεντ Πάτρικ ε, πραγματικά ε, λέμε, ε, καλωσορίζουμε την άνοιξη και λέμε αντίο στο χειμώνα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι σήμερα θα βάλουμε τα θεμέλια μιας καλής προσπάθειας και θα θέσουμε την απαρχή ενός ταξιδιού που θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια από ό,τι φαίνεται και λόγω ε, της θέσης μας ε, στο Κοινοβούλιο με τη συναπόφαση, ανεξάρτητα αν είναι καλό, κακό ή αδιάφορο, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να δούμε ε, τι ακριβώς θα κάνουμε και να είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα αξιοποιήσουμε προς το καλό μας καθώς ε, προχωράμε προς τα μπρος. Πρόεδρε, η προτεραιότητα υπερθμών είναι ο προπολογισμό και το ποσοστό του συνολικού προπολογισμού. Και πρέπει να σα πω ότι με ανησυχεί ιδιαίτερα, διότι κάθε φορά που ε, ακούω τόσου πολλούς να λένε ότι η ΚΑΠ θα έχει λιγότερα, ε, και λιγότερο μερίδιο από τον ε, προπολογισμό τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβω υπόψη ότι από 15 πάμε στα 27 κράτη-μέλη, δεν νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα παίρνουμε ως δεδομένα και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί καθώ θα προχωρήσουμε προ τα μπρος και ω προ τον προπολογισμό. Σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο George Lyon, ο οποίο είπε ότι το μέλλον τη ΚΑΠ θα πρέπει να είναι δίκαιο και για τα καινούργια κράτη-μέλη αλλά και για τα παλιά κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν, τι θέλουμε να πετύχουμε. Εγώ πιστεύω ε, η δίκαιη και φόρο γεωργία που να μπορεί να επιβιώσει και να μπορεί να αντιμετωπίσει τι ε, απαιτήσει που αντιμετωπίζει. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συμβάλλουμε σημαντικά ε, και ε, στο θέμα ε, τη αλλαγή του κλίματο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτέ τι νέε προκλήσει και να τι αξιοποιήσουμε για το συμφέρον μα. Να ε, τι αναπτύξουμε και να κάνουμε ό,τι πρέπει για το μέλλον. Ε, η, η ενιαία πληρωμή ε, είναι κεντρική σημασία για την επιβίωση πολλών γεωργών. Ποιο είναι το μέλλον όμως προς την κατεύθυνση αυτή, είναι ανοιχτό για συζήτηση ε, μέσα στου μήνες. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι, ότι κατά την άποψή μου θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα τις αλλαγές και θα πρέπει να δώσουμε το χρόνο στους γεωργούς για να προσαρμοστούν καταλαβαίνουμε αυτό το οποίο ε, έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ομαλή προσγείωση στο γαλακτοκομικό τομέα. Θυμόμαστε τι έγινε και θυμόμαστε και τι είδου ε, ομαλή προσγείωση ήταν αυτή. Η πρόκληση λοιπόν είναι επίση να αξιοποιήσουμε προ συμφέρον μα και να προσαρμόσουμε τι νέε τεχνολογίε. Δεν μπορούμε ε, να λέμε εμεί όχι και να έρθουν άλλοι και να κυριεύσουν τι αγορέ μα και να φέρουν τα δικά του τρόφιμα. τα οποία παράγονται με άλλα πρότυπα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γεωργοί της Ευρώπης θέλουν να παράγουν καλά τρόφιμα, αλλά δεν θέλουν να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα ε, βάρη λόγω της ε, γραφειοκρατίας. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στις Βρυξέλλες ε, στα, ε, κάθε φορά ε, που υπάρχει μία νέα οδηγία, κάθε φορά που εφαρμόζεται η οδηγία, τι κάνουμε, φέρνουμε περισσότερη γραφειοκρατία στους γεωργούς και αυτό κατά την άποψή μου είναι ένα από τα μεγαλύτερα σφάλματα που διαπράττουμε και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να φύγουμε από αυτήν την κατάσταση. Έχουμε τώρα την ευκαιρία να θέσουμε το εξή ερώτημα. Τι θέλουμε. Θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε το ανέφερε στη δική του έκθεση και ο Τζόρτζ. Θέλουμε τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2 η διαμόρφωση ε, είναι, ε, αποτελεί ε, μέρος του μέλλοντος. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Και πραγματικά νομίζω ότι αν δεν κάνουμε κάτι προς την κατεύθυνση αυτή, εμείς ποιος θα το κάνει. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα σημεία αυτά και να σημειώσουμε πρόοδο, γιατί σε τελευταία ανάλυση, όταν ο Φρας Φίσλερ ε, έφερε τη διαμόρφωση, έφερε τον, το πυλώνα 2. Ε, δεν πρόβλεψε όμω τα κονδύλια για την υποστήριξη ε, τη κοινότητα των Γεωργών, παρόλο που ήταν ευχή πρόθεση κάτι τέτοιο. Ε, αυτό ήταν το αδύνατο σημείο. Τελειώνω ε, και καταλαβαίνω, Πρόεδρε, θα ανυπομονείτε να σταματήσω. Αλλά να σα πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση. Εάν η συγχρηματοδότηση ε, δεν ε, αφορά ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε υπάρχει ο κίνδυνο να μετακινηθούμε από την κοινή αγροτική πολιτική η οποία θα πάψει να υπάρχει ε, ως ε, κοινή αγροτική πολιτική. Ε, θα πρέπει να, να θέσουμε το ξερότημα στον εαυτό μας. Έχουμε αρκετά εργαλεία. Η απάντηση είναι όχι. Πρέπει λοιπόν να βρούμε αυτά τα νέα εργαλεία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ε, πρέπει, ε, έχουμε να κάνουμε πολλά και δεν θα πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Ε, γιατί πρέπει, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον της γεωργίας, για το μέλλον των γεωργών. Θα πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στην κοινότητα της υπαίθρου. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μας δίνουν τρόφιμα στο μέλλον. Και αυτοί είναι οι άνθρωποι που κατά την άποψή μου θα μπορέσουν να συμβάλλουν ιδιαίτερα σε αυτό το οποίο ε, απαιτεί η σημερινή κατάσταση, λαμβάνοντα υπόψη την αλλαγή του κλίματο κτλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, James. Και τώρα δώσω το λόγο στον George Lyon με την ιδιότητά του του εισηγητή. Ε, όχι, συγγνώμη, του εκπροσώπου των φιλελευθέρων και όχι με την ιδιότητά του του εισηγητή. Θα είμαι πολύ στομός γιατί θα μπορούσα να συνοψίσω και στο τέλος. Από αυτά που ακούω εγώ από τους ε, παρεμβαίνοντες είναι ότι η οικονομική κρίση και οι περιβαλλοντικές, οι κλιματικές αλλαγές καλύτερα είναι οι κύριοι παράγοντες ε, που καθοδηγούν οποιασδήποτε εξελίξεις στην ε, γεωργία και που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Από εκεί και πέρα συγχρηματοδότηση από την πίσω πόρτα μην με επανεθνικοποίηση και δεν θα πρέπει να την υποστηρίξουμε, ε, η σταθερότητα η προβλεψιμότητα στην πολιτική μας είναι απαραίτητη όρη οι εκπρόσωποι των γεωργών μας λένε, νομίζω ξεκάθαρα με τους εκπροσώπους τους, δεν φοβούμαστε την αλλαγή, αλλά να ξέρουμε που πάμε, να έχουμε μια σταθερότητα και προβλεψιμότητα, ώστε να ξέρουμε ότι μπορούμε να προσαρμοστούμε στους νέους στόχους. Αυτά είναι πιστεύω κυρίως τα συμπεράσματα από τις παρατηρήσεις τους, να δώσουμε τη δυνατότητα στους γεωργούς να βλέπουν το μέλλον μπροστά τους, να υπάρχει ε, η ευκαιρία και για τους νέους να μπουν στο επάγγελμα του γεωργού και να βλέπουν το, το μέλλον τους αίσιο. Αυτά νομίζω ακούγονται πάνω κάτω από τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν από τους Γιώργους. Περισσότερη υποστήριξη δεν ζητούν. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο των Πρεσίνων, ο Μάρτιν Χόσλινγκ. Κυρίε και κύριοι, καταρχάς ευχαριστώ τον George Λάιον και για την ευκαιρία που μας δίνει, αλλά και τους ομιλητές. Ήταν πολύ σημαντικό το θέμα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια σημεία. Ο George Lyon είπε την προηγούμενη φορά ότι για την έκθεσή του προβλέπει τον ε, στόχο μιας πράσινης κάπου που χρειαζόμαστε. Σε αυτό φυσικά απερίφραστα προσυπογράφω. Και θα πρέπει, πιστεύω, η κοινή γεωργική πολιτική να γίνει πιο οικολογική. Κάποιοι από τους ομιλητές επίσης ε, είπαν ότι θέλουν περισσότερη ότι έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο από ότι στο Συμβούλιο θα δούμε στο τέλος όλη αυτή τη συζήτηση αν έχουν δίκιο. Νομίζω όμως ότι πρέπει η συζήτηση, ο διάλογος να αναπτυχθεί στο δυνατόν σε πιο ευρύ όρους, όχι μόνο μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά ευρύτερα, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο με βάση αυτό που εννοεί και ο Γεωργός και όλος ο κόσμος, να ξέρουμε τι σημαίνει ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική σε αντιπαράθεση με μια άλλη γεωργική πολιτική. Επίσης, στη στρατηγική 2020 ακούστηκε, αναφέρθηκαν κάποιοι όροι, πολύ όμως ε, περιθωριακά ε, για την κοινή γεωργική πολιτική και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να μην παραγνωριστεί ο ρόλος της ως κεντρικής κοινή πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να υπογραμμίσουμε ότι χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργική πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι εδώ στην Επιτροπή μας. Ωστόσο δεν είναι όλα ρόδινα στην κοινή γεωργική πολιτική όπως την είχαμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν αρκετές επικρίσεις, επικρίσεις που έχουν να κάνουν και με την κατανομή των χρηματοδοτικών μέσων, με την ανισότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επικρατεί μεταξύ τόσο κρατών μελών όσο και διαφόρων ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων ή γεωργών και θα πρέπει να δούμε τελικά ποιος επωφελείται από τα διατηθέμενα κονδύλια, πού πάνε τελικά τα λεφτά που δίνουμε. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε. Και επίσης κοινή γεωρική πολιτική σημαίνει ταυτόχρονα ότι δεν έχουμε μπορέσει να προσαρμόσουμε το εισόδημα των γεωργών στους στόχους που είχαμε ορίσει, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα και ο γεωργός να υποφεληθεί από μια αύξηση των τιμών, να ενισχύει το εισόδημά του όταν η αγορά πάει καλά. Αυτό Επισημάνθηκε ήδη ότι η λύση θα δοθεί στο πρόβλημα του σωτήματος των γεωργών μέσα από μια άλλη γεωργική πολιτική, άλλη αγορά γεωργική. Έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία μεταξύ του, κόστος, του κόστους ε, παραγωγής ενός προϊόντος και της τιμής που πληρώνει τελικά ο καταναλωτής τον το αγοράζει. Ταυτόχρονα για την Βία Καμπεσίνα θα ήθελα να επισημάνω ότι πολύ σημαντικό βρήκα αυτό που μας εξέφρασε ο πρόσωπός της, δηλαδή την ε, ευθύνη που φέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεν ε, είναι δυνατόν να έχουμε ρυθμίσεις οι οποίες στρεβλώνουν την αγορά και οι οποίες με τις επιδοτήσεις εξαγωγών φέρνουν σε δυσμενέστερη θέση ή ε, μετατρέπουν σε θύματα ενός αθέμητου ανταγωνισμού τους μικρούς παραγωγούς στις αναπτυσσόμενες χώρες. Χρειάζεται λοιπόν μια διαφορετική λύση για τα προβλήματα αυτά. Ένα νέο σύστημα το οποίο πιστεύω θα μπορέσει να συμβάλλει και στην διαφύλαξη των μικρών παραγωγών, στην διατήρηση των μικρών ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων και στα τρίτα κράτη, στα αναπτυσσόμενα κράτη. Ταυτόχρονα θα πρέπει μια νέα γεωργική πολιτική να συμπεριλαμβάνει στους, ε, στους στόχους της και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και την ε, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Αυτό πρέπει να είναι ένας στόχος σαφής στη νέα γεωργική πολιτική μας. Για το δημοσιονομικό πλαίσιο, πιστεύω, θα πρέπει να τοποθετηθούμε όταν θα έχουμε συγκεκριμένο ε, ιδέα για το περιεχόμενο των στόχων που θα ορίσουμε και ανεξαρτήτως αυτών θα πρέπει να γνωρίζουμε για να διαμορφώσουμε τους στόχους θα πρέπει να γνωρίζουμε να έχουμε ξεκαθαρίσει τι θέλουμε ως ιωρική πολιτική. Θέλουμε και να διαφυλάσει την ύπεθρο, θέλουμε να διαφυλάσει το τοπίο μας και με αυτό νομίζω μπορούμε να εξασφαλίσουμε, με σαφεί στόχου μπορούμε να εξασφαλίσουμε για την υποστήριξη τη κοινή γνώμη. Γιατί δεν νομίζω ότι η κοινή γνώμη στέκεται αρνητικά απέναντι στην κοινή γεωργική πολιτική. Υπάρχουν οι επικρίσει, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι παραγνωρίζει κανεί τη σημασία τη γεωργία στην Ευρώπη. Έχουμε συζητήσει επί μακρόν τα θέματα αυτά. Εμεί ω Κοινοβούλιο ασφαλώ όλη αυτή την ε, συζήτηση θα την αξιοποιήσουμε στο μέγιστο. Ήταν ε, πολύ καλό ο διάλογο και πιστεύω ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί και περαιτέρω διάλογο, ευρύτερο διάλογο και μέσα από ε, όλο, τον κόσμο της γεωργίας για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η εκπρόσωπος ε, της ε, Γκουέι ο εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ, ο κύριος Λεϊερικ Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές και τον εισηγητή. Θέλω να πω το εξή. Εμείς εδώ λέμε πολλές γενικολογίες και θέτουμε πολλούς κοινού στόχους, γενικούς στόχους, που είναι σωστοί. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν απαραίτητο να εμβαθύνουμε σε ορισμένα ζητήματα, γιατί αλλιώς οι γενικοί μας στόχοι δεν έχουν καμία ευκαιρία να καταλήξουν σε τίποτα. Λέμε πολλές φορές ότι η ΚΑΠ εκπλήρωσε συνολικά την αποστολή της. Ναι, μακροοικονομικά και όσον αφορά στην τροφιμική αυτάρκεια, ναι. Αλλά η κατάσταση του μικρομεσαίου αγρότη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι δραματική και αυτό ξεχνάμε να το πούμε. Ε, ε, ε, υπόκειται σε μια τεράστια μείωση εισοδήματος, χρέωση, πτώχευση και τελικά κόσμος ο οποίος εξαφανίζεται γιατί είναι αναγκάζεται να κλείσει τη γεωργική του εκμετάλλευση στην Γαλλία. Πολλοί αγρότες ε, όχι μόνο οι μικροί αγρότες ε, ε, γράφονται στα, διάφορα ταμεία για να πάρουν την ελάχιστη, το, επίδομα, το, το επίδομα επιβίωσης. Νομίζω λοιπόν ότι η εκπλήρωση των στόχων τουλάχιστον σε επίπεδο βιωτικού επίπεδου δεν είναι αλήθεια. Επίσης θα πρέπει να συζητήσουμε τι τύπου γεωργία χρειαζόμαστε να είναι αποτελεσματική και κοινωνικά αλλά και οικονομικά. Υπάρχει διαφορά στο να θέλουμε μια γεωργία που να βασίζεται στους αγρότες και μια γεωργία βιομηχανικού τύπου στα πλαίσια του ανταγωνισμού η μείωση των τιμών που έχουμε σήμερα γιατί έχουν ληφθεί πολιτικές αποφάσεις δεν είναι το Άγιο Πνεύμα που οδήγησε στη μείωση των τιμών. Πολιτικές αποφάσεις οδήγησαν στην απορρίθμιση των τιμών και στην εντατικοποίηση της παραγωγής, αύξηση της παραγωγικότητας με πολύ σημαντικά στρεβλά φαινόμενα. Αυτό είναι αντίθετο με την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά και οι δασμοί και η, η, και η κοινωνική προτίμηση. Ε, αν εμείς συνεχίσουμε όπως ε, σήμερα, δηλαδή να εισάγουμε γεωργικές ε, παραγωγές και τρόφιμα σε πολύ χαμηλές τιμές από τρίτες χώρες, εμποδίζοντάς τις να είναι ίδιες αυτάρκεις και να, και να είναι και ανταγωνιστικές απέναντί μας, τότε τι κάνουμε. Εμείς ε, δεν λύνουμε ούτε το πρόβλημα του λοιμού και εξαφανίζουμε τους αγρότες μας. Το θέμα λοιπόν ε, της, του να βρεθεί ένα σύστημα ε, κοινή γεωργικής πολιτικής συνδυασμένο και με την κοινωνική διασφάλιση των δικών μας αγροτών και με έναν σωστό ανταγωνισμό χρειάζεται για το θέμα τώρα των ενισχύσεων, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να, υπάρχει, να υπάρχουν όροι για τη χορήγηση αυτών των ενισχύσεων, ούτως ώστε να ευνοήσουμε την κοινωνική προόδο και το περιβάλλον. Δεν βάζουμε επίσης ποτέ το ζήτημα των ενδοευρωπαϊκών μας σχέσεων. Βρισκόμαστε εμεί σε ένα σύστημα το οποίο οδηγεί στον ανταγωνισμό των Ευρωπαίων αγροτών μεταξύ τους. Γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς, ας πούμε, στη φάση της ε, παραγωγής ε, φρούτων και λαχανικών, να έχουμε ένα ημερολόγιο, ένα χρονοδιάγραμμα ε, εισαγωγών συντονισμένο, διότι τελικά είναι οι έμποροι και οι μεσάζοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Είναι κατά μιας αλληλέγγυας Ευρώπης αλλά είναι συμβατό με την αρχή του ανταγωνισμού που στρεβλώνει πολλά πράγματα. Μιλάμε για αυτάρκεια. Σε ορισμένες χώρες όμως υπάρχουν παραγωγές όπου δεν υπάρχει αυτάρκεια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το αρνήσιο κρέας και για το βοδινό. Δεν είμαστε αυτάρκοι. Προτιμούμε να εισάγουμε ε, από άλλες χώρες, παράδειγμα προβατήσιο κρέας. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ρίχνει την ιδέα ενός σχεδίου πρωτεΐνης για την ίδια, αντί να εισάγει πρωτεΐνες όπως το κάνουμε σήμερα, πρωτεΐνες με βάση, που εισάγουμε πρωτεΐνες με βάση γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Σίγουρα ο Γιώργος ο αγρότης έχει μία αποστολή κοινή ωφέλεια και το γεγονός παραγωγής πρώτων γεωργικών υλών θα πρέπει να θεωρείται ένα κοινό αγαθό. Αλλά με αυτούς τους όρους αυτό είναι σύμβατο με τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων στην ΠΟΕ όπου θεωρούμε τις γεωργικές πρώτες ύλες ως εμπορεύματα και όχι ως κοινό αγαθό και αυτό με όλες τις επιπτώσεις. Ε, εγώ είμαι κοντά σε αυτήν την άποψη των φίλων μας ε, της Βία Καμπεσίνα μία κάπη που να έχει ε, πολλαπλούς ρόλους σας ευχαριστώ. Πριν συνεχίσουμε, δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της ΟΚΕ, τον κύριο Λουίς Ρίμπε, ο οποίος είναι εισηγητής για τη γνωμοδότηση για το μέλλον της ΚΑΠ. Κύριε Ρίμπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε που μας επιτρέπεται να λάβουμε το λόγο εδώ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και θα ήθελα να εκφράσω και την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι έχει καθοριστικά πλέον και καθοριστικές και νέες εξουσίες στο θέμα τη Γεωργίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορεί έτσι να γίνει μια συζήτηση όπου οι εκπρόσωποι των πολιτών και τα κόμματα που τους, ε, στα οποία ανήκουν θα έρθουν σε αντιπαράθεση απόψεων για να συστήσουν τα θέματα αυτά. Θέλω να σημειώσω ότι και εμεί έχουμε μια γνωμοδότηση και ελπίζουμε ότι αύριο με την έγκρισή τη ε, θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στι εργασίε σα. Τους ε, τελευταίους μήνες έγινε λιγότερη συζήτηση για τους στόχους τους οποίους θα πρέπει να επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερο για τα μέσα έγινε συζήτηση, δηλαδή για τα κονδύλια και για το πώς θα κατανέμονται. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει περισσότερο να δώσουμε την έμφαση στους στόχους. Αυτές είναι οι νέες προκλήσεις, όπως άλλωστε αναφέρθηκαν και νωρίτερα, οι κλιματικές αλλαγές. Και επιτρέψτε μου εδώ η προστασία από τις κλιματικές αλλαγές. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είναι βιοπικιλότητα θα πρέπει και αυτή να τη συστήσουμε στους στόχους, διότι η γεωργία συμβάλλει ιδιαίτερως στη διαφύλαξη της, δια... της ε, μας ή μπορεί να οδηγήσει και στο τέτοιο αποτέλεσμα, εάν δεν έχει σωστή λειτουργία. Επίσης, λοιπόν, από πλευρά Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής θα θέλαμε να πούμε ότι το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο θα πρέπει να αποτελέσει ένα... θα πρέπει να έχει ένα ε, θα πρέπει να είναι το περίγραμμα της κοινή γεωργικής μας πολιτικής το light build όπως θα λέγαμε, θα πρέπει να έχουμε μια πολύ λειτουργικότητα της ε, γεωργίας, να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη ψαλίδα που όλο και ανοίγει στην καθημερινή ζωή, γιατί το γεωργικό μοντέλο, μοντέλο της Ευρώπης ε, υφίσταται σημαντικές πιέσεις από τις αγορές για την μείωση των τιμών ή τις, διακυμε... τις κειμενόμενες δαρκοστιμές, την ανάγκη για προσαρμογή σε νέες συνθήκες, για ε, εξειδίκευση των εκμεταλλεύσεων, για εξορθολογισμό για συγκέντρωση σε ορισμένες περιοχές, για να αναφέρω ως παράδειγμα τις παράκτιες περιοχές που αναφέρθηκαν και νωρίτερα. Από τη μία πλευρά συγκέντρωση λοιπόν σε ορισμένες ζώνες, από την άλλη ε, απερίμωση ορισμένων ζωνών ή περιοχών. Νέες λοιπόν συνθήκες οι οποίες πιέζουν και απειλούν τη γεωργία μας. Και γι' αυτό σας παρακαλούμε την πολιτική που θα χαράξετε να τη χαράξετε για αυτό το ευρωπαϊκό μοντέλο της γεωργίας. Δηλαδή Χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση με βάση τους στόχους, με γνώμονα τους στόχους. Η γεωργική πολιτική δεν μπορεί να χαραχθεί μόνο με γνώμονα την αγορά ή τις τιμές. Πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε ως μοντέλο. Τι στόχους θέλουμε να επιτελεί αυτό το μοντέλο. Και τότε θα του διαθέσουμε και τα μέσα που χρειάζεται για να έχουμε μια συνεπή πολιτική, μια συνεκτική πολιτική και με πολύ μεγάλη χαρά άκουσα σήμερα ότι οι συνέπειες της απορρίθμισης ε, επισημάνθηκαν ως ένας από τους κύριους λόγους που οδηγούν σε προβλήματα την ε, γεωργική πολιτική. Η αποσταθεροποίηση των αγορών επίσης. Άρα θα πρέπει έναν από τους στόχους που θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ως στόχους ευρωπαϊκής πολιτικής ε, να εντοπίσουμε τη σταθεροποίηση των αγορών, το σταθεροποιητικό ρόλο της κοινωνικής πολιτικής ως προς τις αγορές, μετά τη Λισαβόνα ιδιαίτερα ως στόχο της Λισαβόνα πρέπει να το εντοπίσουμε και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η συζήτηση, ο διάλογος που θα αναπτυχθεί και θα ακούσουν ασφαλών και άλλα ζητήματα ως προς τα μέσα λοιπόν που θα έχει η Γεωργία θα πρέπει να περιλάβει και τη διάστασή της σταθεροποίηση των αγορών. Επίσης, η γεωργική πολιτική δεν είναι μόνο ανοίγω το πορτοφόλι και δίνω χρήμα έχει άλλα μέσα, έχει πολύ περισσότερα μέσα από τη διάθεση κονδυλίων η γεωργική πολιτική. Δεν πρέπει να περιοριστούμε μόνο στην αντιπαράθεση απόψεων ως προς το, ε, τα κονδύλια. Εμείς λέμε ναι για το μέλλον, διατήρηση των ε, πληρωμών, των ενισχύσεων, αλλά με ένα άλλο μοντέλο σιγά σιγά. είχαν κάποιο λόγο ύπαρξη αυτέ οι πληρωμέ, όταν το 1992 είχαμε σημαντική πτώση των τιμών, παραδείγματι, και θα πρέπει να εξυπηρετούν κάποιο στόχο αυτέ οι ενισχύσει όπου χρειάζονται. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει αυτές να είναι σε σύζευξη με κάποιον στόχο. Δεν μπορεί κάποιο να πάρει ένα αεροπλάνο και να, ανοίξει ε, από την πόρτα του αεροπλάνου να πετάει χρήμα πάνω από την Ευρώπη, πάνω από τα χωράφια τη Ευρώπη και να πούμε αυτό αρκεί. Πρέπει το χρήμα που θα διατίθεται να εξυπηρετεί και το στόχο της προστασίας των ζώων και το στόχο της ε, διαφύλαξης της υπαίθρου μας, της καλής παραγωγής. Όλους αυτούς τους στόχους λοιπόν θα προσδιοριστούν με τη συζήτηση που θα αναπτυχθεί. Επίση, θα πρέπει να διαφυλαχθούν οι γεωργικέ εκμεταλλεύσει. Θα δούμε με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί αυτό ο στόχο. Πάντω, δεν θα πρέπει να υπάρξει κατά αποκοπή ενιαία πρημοδότηση επιφάνειας, αυτό είναι αδικαιολόγητο, θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση, είτε πρόκειται για γεωργική εκμετάλλευση, δηλαδή για ε, χωράφι, είτε πρόκειται για κτηνοτροφική εκμετάλλευση. και άλλωστε έχουμε και αντίστοιχε παρατηρήσει εμεί μέχρι την έκθεσή μα, που θα εκρεθεί όπω σα είπα την Ολομέλεια. Ε, οπότε θα μπορείτε να δείτε τι παρατηρήσει μα. Επίση, θα ήθελα να πω ότι πρέπει να έχουμε συνέπεια, συνοχή στι ε, επενδύσεις, ενίσχυση των επενδύσεων για τη γεωργία και τι γεωργικές εκμεταλλεύσεις με στόχο πάντα την ε, προαγωγή και διαφύλαξη του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου και όχι την εκβιομηχάνηση της γεωργίας μας. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ε, ξέρω ότι είναι μια διαδικασία μακροχρόνια, θα διαρκέσει τουλάχιστον 2-3 χρόνια, αλλά πιστεύω ότι θα καταλήξει πολύ καλά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την ε, ΕΟΚΕ. Και τώρα ας ξεκινήσουμε με τις ε, ε, παρεμβάσεις μέχρι τις 5, 5 και 5. Για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα μιλήσουν μετά τους εμπειρογνώμονε. Κύριε Παπαστάμκος, ο πρώτος ομιλητής. Θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά για τη διοργάνωση αυτή τη δημόσια ακρόαση, όπω επίση θα ήθελα να ευχαριστήσω του συγητές για τι παρεμβάσει του, για τι γόνιμε και δημιουργικέ παρεμβάσει του, τον κύριο Χανιώτη για την οικονομική αναλυτική του παρέμβαση, καθώς και τους ε, εκπροσώπους των ε, αντιπροσωπευτικών φορέων για τις ε, διαφορετικές ματιές του Ευρωπαϊκού Νότου, της Κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης ή του Ενωμένου Βασιλείου στο μείζον θέμα της αναθεώρησης της ΚΑΠ, της μετά το 2013. Δεν θα επεκταθώ σήμερα, γιατί το έκανα σε προηγούμενη συνεδρίασή μας, στη δικιά μου μείζωνα προσέγγιση ως προς την ΚΑΠ μετά το 2013, αλλά θα αρκεστώ σε μερικές αντανακλαστικές παρατηρήσεις. Κύριε Πρόεδρε, η Κομισιόν έχει την νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά συγχρόνως είναι και ένα σώμα τεχνογνωσίας. Εμείς είμαστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ένα πολιτικό σώμα, βεβαίως και συνομοθετικό σώμα μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει το εξουδετικό θεμέλιο, την αρμοδιότητα να έχουμε μια ουσιαστική κανονιστική παρέμβαση. Εγώ θα έλεγα στον κύριο Λάιον, στον εισηγητή μας, αλλά είναι και ευθύνη όλων ημών, που είμαστε φορείς της ε, ευθύνης δημοκρατικής λογοδοσίας απέναντι στο εκλογικό μας σώμα, στην Ευρωπαϊκή Ήπεθρο, να κωδικοποιήσουμε πολιτικά τη δικιά μας προσέγγιση, τις δικές μας θέσεις για την ΚΑΠ μετά το 2013. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν δεν θα κάνει τη δουλειά της, δεν θα εκπονήσει την ε, δικιά της πρόταση, αλλά ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως πολιτικό σώμα, καλούμαστε και είναι ευκαιρία αυτή να διατυπώσουμε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών και θέσεων συμπεφωνημένα εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας και με αυτό να απευθυνθούμε προς την Επιτροπή αλλά και στο άλλο πόλο της νομοθετικής διαδικασίας. Κατά τη γνώμη μου προτεραιότητα δεν πρέπει να είναι ο προϋπολογισμός. Αντίθετα, ανάστροφα, προτεραιότητα πρέπει να είναι το ποιο, ποια κοινή αγροτική πολιτική θέλουμε να οικοδομήσουμε και μετά να, έρθουν, να έρθει η δημοσιονομική πλαισίωση αυτού του μοντέλου που θα αποφασίσουμε, θα συναποφασίσουμε. Ο πρώτος πυλώνας, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, τεκμηριώνει, υποβαρθρώνει αυτό που λέμε κοινή αγροτική πολιτική. Δεν, το, δεν συζητούμε για κατάργηση του πρώτου ε, πυλώνα έγιναν αναφορές στο αγροτικό εισόδημα και χάρηκα που άκουσα τον κύριο Σον Λάιτερ να αναφέρει ε, ποσοτικά στοιχεία ότι το εισόδημα του, το μέσο αγροτικό εισόδημα είναι πολύ χαμηλότερο από το μέσο εργατικό ε, μισθό. Όπως επίσης και ο δικός μας αναπληρωτής ε, συντονιστής, ο κ. Νταντέ, αναφέρθηκε στις προδιαγραφές παραγωγής. Γνωρίζω ότι η Γαλλία και ορθώς αυτό τον αγορεύει σε κορυφαία προτεραιότητα δεν υπάρχουν οι ευφυείς, οι λιγότερο ελαστικοί, οι περισσότερο αυστηροί στην παγκόσμια στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Εξαιρώ βεβαίω τα LDCs, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ομοιομορφία ή σε ισοδυναμία προδιαγραφών παραγωγής. Δεν μπορούμε να έχουμε με άλλους όρους ασφάλειας τροφίμων να, να τα εισαγόμενα από ότι τα εγχωρίως τα ευρωπαϊκώς ε, παραγόμενα. Άκουσα τη λέξη προστατευτισμός από τον κύριο Κένταλ. Κοιτάξτε, μιλούμε για δημόσια αγαθά. Τα δημόσια αγαθά, η παραγωγή τους, χρειάζονται δημόσια, ενώ ευρωπαϊκή, χρηματοδότηση. Τα δημόσια αγαθά και η διατροφική κυριαρχία δεν μπορούν να αφήνονται στις τύχες των αγορών. Μην γελιόμαστε. Είδαμε ότι ο πιο προβλημένος τομέας που αφέθηκε στην τύχη των αγορών, ο χρηματοπιστωτικός, είδαμε πού οδήγησε την παγκόσμια ε, χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική. Και επειδή μιλούμε για, και για προϋπολογισμό, θέλω να πω να μην παραβλέπουμε ότι, και τελειώνω με δύο παρατηρήσεις, προτελευταία είναι αυτή, ότι η ποσοστιαία συμβολή της κοινή αγροτικής πολιτικής στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ είναι μεγαλύτερη από την επιβάρυνση του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Και αυτό πρέπει να είναι επιχείρημα το οποίο να το προτάσουμε έναντι όσων μιλούν για την ανάγκη περικοπών. Και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Έχω την αίσθηση ότι τόσο η νέα στελέχωση της Κομισιόν, αλλά όσο και εμείς, και ορθώς βέβαια σε ένα σημείο, αποδίδουν μεγάλη προτεραιότητα στην οργάνωση τα του οίκου μας, όπως είπε και ο Επίτροπος, στην εσωτερική οργάνωση της κοινή αγροτικής πολιτικής διαγράφεται ένας κίνδυνος και θέλω να τον καταστήσω σαφή αυτόν τον κίνδυνο. Να προέλθει αναθεώρηση κοινή αγροτικής πολιτικής εκ των έξω ή εκ των άνω στο, στις διαπραγματεύσεις του γύρου ε, της Δόχα. Και αυτό πρέπει να το έχουμε ε, πάνω στην ατζέντα μας καθημερινά. Οπότε θα έρθει μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας πει «Α, τώρα πρέπει να συμμορφωθούμε με το διαπραγματευτικό αποτέλεσμα του γύρου της Δόχα». Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Παπαστάμκο και συνεχίζουμε με τις ε, παρεμβάσεις ε, με τον επόμενο μιλτή. Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Καπούλα Σάντος έχει απόλυτο δίκιο. Χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση στην γεωργική πολιτική. και νομίζω ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ως, τόσο συχνά ε, τη λέξη ανταγωνιστικότητα. Ήμουν πέρυσι στην Ιαπωνία και μπόρεσα να δω ότι ε, παντού ε, καλλιεργούν ρύζι. Δεν ξέρω πώς φυτρώνει το ρύζι αυτό, αλλά φυτρώνει παντού. Και μπορεί κανείς να αγοράσει, όμως ταυτόχρονα, δίπλα είναι η Κίνα που είναι πολύ φτηνότερο το, το ρύζι. Και όμως η χώρα αυτή γνωρίζει το πόσο σημαντική είναι η διατροφική ασφάλεια. Ε, και διαθέτει και, και φαντασία η Ιαπωνία. Και η Ευρώπη πέστη πολλά, αλλά δεν διαθέτει φαντασία. Αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια είναι μια εκποίηση της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ε, και βλέπουμε τι ε, επιπτώσει έχει αυτό στην παραγωγή. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα έναντι των άλλων, των ΙΠΑ, τη Βραζιλία κτλ. Με βάση διάφορα πρότυπα, ανοιχτή αγορά κτλ. Και ο κύριο Κάντελ αναφέρθηκε στο ζήτημα αυτό, Κένταλ αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Άρα λοιπόν, για τη λέξη ανταγωνιστικότητα, να χρησιμοποιούμε την επιβίωση, τη λέξη επιβίωση. Η, η Ευρωπαϊκή Γεωργία προσπαθεί να επιβιώσει για καλύτερου καιρού που θα έρχουν. Και αυτό το ακούσαμε και από άλλου ομιλητέ. Ε, θα έρθουν οι καλύτεροι καιροί. Γιατί έχουμε και περισσότερες εκτάσεις για να καλλιεργήσουμε άρα, ε, τώρα. Άρα θα πρέπει ε, να φροντίσουμε τη γεωργία. Και μην ξεχνάτε στο μέλλον τα, τα τρόφιμα θα αποκτήσουν στρατηγική σημασία. Επίσης, ε, το θέμα των, ε, της ίσης αμοιβής, ε, χαίρομαι που το έθιξε ο, ο συνάδελφος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Και όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για μετά από το 2013. Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται στα 600 το εκτάριο και άλλες ε, όπω η Πολωνία, βρίσκεται στα 100 το εκτάριο. Και άλλες ακόμα, όπω η Λετωνία, που είναι ακόμα πιο χαμηλά. Άρα λοιπόν ε, ε, έχουμε διαφορές όχι μόνο ανάμεσα στα παλιά και στα καινούργια μέλη, ανάμεσα και στα παλιά. Πρέπει λοιπόν να δούμε το ζήτημα αυτό. Και ε, ξέρω τι ε, γίνεται στις χώρες που αυτές που έχουν υποστεί η διακριτική μεταχείριση. Δεν θα συμφωνήσουν, για παράδειγμα στη χώρα μου, οι Γεωργοί δεν θα, συμφωνήσουν με την συνέχεια αυτών των διαφορών. Δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Τι θα κάνουμε λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των διαφορών. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα πείτε παίρνουμε από αυτούς που παίρνουν περισσότερα. Γιατί άμα πάρουμε από αυτού που παίρνουν περισσότερα, τότε και εκεί θα είναι τεράστιε οι αντιθέσει. Άρα λοιπόν έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δημοσιονομικό πρόβλημα για την κοινή αγροτική πολιτική. Αλλά και ε, πρόβλημα ε, όσον αφορά τον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Έχουμε και τη συνθήκη τη Λισαβόνα τώρα. Μα σα λέω ότι πέρυσι, όταν συζητήσαμε τη συνθήκη τη Λισαβόνα, υπήρχε έτσι ένα πνεύμα ενθουσιώδες και ε, πρέπει να σας πω ότι όταν τους ε, ρωτούσαμε ε, γιατί την πρώτη φορά δεν δεχόσασταν τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Ε, στη συνέχεια είχαμε, ε, δεν ακούσαμε κάποια απάντηση. Μετά ε, είχαμε ε, και, το, και τον Πολωνό πρόεδρο, ε, τον πρόεδρο τη Τσεχία που δίστασαν να υπογράψουν. Υπήρξε και μια δυσαρέσκεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλο πάντων τελικά υπογράφηκε η συνθήκη Λισαβόνα. Η συνθήκη της Λισαβόνας. Και τώρα τι γίνεται. Ε, υπάρχει ένα είδο εγωιστική τάση, όπου κανένα δεν θέλει να πληρώσει αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσει. ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, λιγότερο από, λιγότερο από το 1% του ΑΕΠ. Μα καταλαβαίνετε ότι ε, λαμβάνοντα υπόψη τι δαπάνε, είναι πολύ άνηση η κατάσταση. Αν δεν έχουμε ένα πιο σωστό προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιλύσουμε τις, ε, τα προβλήματά μα, δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει και δεν πρόκειται να έχουμε αποκατάσταση δικαιοσύνη προ την κατεύθυνση αυτή. Εάν θέλουμε να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ μας, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε την, ε, ε, τα αποτελέσματά μας, τότε χρειαζόμαστε δικαιοσύνη ε, και όχι το αντίστροφο. Χρειαζόμαστε λοιπόν κονδύλια για ασφάλεια που είναι πολύ σημαντική σε συγκεκριμένο τομέα. E Η κυρία Γέγκε μετά ο, ο Ζωσέ Μποβέ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, η ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική είναι μέχρι στιγμή η μόνη κοινοτικοποιημένη πολιτική. Αυτό ήθελα να το δηλώσω προκαταβολικά. Ε, όταν λοιπόν ε, συζητούμε αυτήν την κοινή γεωργική πολιτική, τη μόνη κοινοτικοποιημένη, και το, τα μοντέλα της, θα ήθελα εγώ να σημειώσω ότι πρόκειται για ένα μοντέλο, ναι, το οποίο έχει πολλά χρόνια ιστορία στην πλάτη του, έχει μειονεκτήματα, αλλά από την άλλη αν εξετάσουμε όλη του την ιστορία, τι μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει ένα καλό περιβάλλον, ένα καλό τοπίο, καθαρό τοπίο, πράσινο περιβάλλον, καθαρό περιβάλλον. Ο γεωργός μας, ο κυπουρός, ο κτηνοτρόφος έχουν κάνει καλή δουλειά. Πάνω απ' όλα με αυτή τη βάση πρέπει να ξεκινούμε. Μια καλή δουλειά και θέλουμε να συνεχίσουν να κάνουν καλή δουλειά. Γι' αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ. Διότι δεν είμαστε εμεί οι υπέτειοι αυτή τη οικονομική κρίση, ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε σε ολόκληρο τον κόσμο. Όμω μα πλήττει η οικονομική κρίση. Ο κοινοτικό προπολογισμό μα λένε έχει, ε, δίνει μεγάλο μερίδιο του στην γεωργία. Ναι, όμω είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση τη γεωργία για να μπορέσει να συνεχίσει να επιτελεί το έργο τη και στο μέλλον. Ο κύριος Λάιον είπε ότι 50% του ε, γεωργικού εισοδήματος προέρχεται από τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, δηλαδή από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Ναι, αλλά αν θέλουμε να έχουμε καλή προστασία των ζώων, αν θέλουμε να έχουμε υψηλέ προδιαγραφέ παραγωγή, υψηλή ποιότητα και ασφάλεια τροφίμων, εάν θέλουμε να έχουμε επιστηστική ασφάλεια και αυτάρκεια, πρέπει να διαθέσουμε τα χρήματα αυτά. Και όντω, οι στόχοι των νέων κλίσεων που έχουμε μπροστά μας πρέπει να προσδιοριστούν. Ο κύριο Λάιον έχει μια καλή βάση εργασία, πιστεύω ένα καλό έγγραφο εργασία υποβάλλει και Χάρη σε αυτό θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ όλους εκείνους οι οποίοι σήμερα είπαν ότι χρειαζόμαστε μια κοινή γεωρική πολιτική, γιατί κανείς δεν υποστήριξε την επανεθνικοποίηση, πράγμα το οποίο σε προηγούμενες συζητήσεις είδα να συμβαίνει, δηλαδή ακούσαμε σε άλλες συστήσεις διαφορετικούς τόνους και στόχους. Σήμερα όμως λέμε ότι θέλουμε μια κοινή γεωρική πολιτική και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για το στόχο και της οικολογίας και των κοινωνικών προδιαγραφών, αλλά Χρειαζόμαστε και την αποτελεσματικότητα και την οικονομία, την οικονομική απόδοση δηλαδή και την καινοτομία στη γεωργία μας. Και αυτοί είναι οι στόχοι για τους οποίους πρώτα απ' όλα πρέπει να αγωνιστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Ελίζαμπεθ. Ο κύριος Μποβέ. Έχει το λόγο και μετά συνεχίζουμε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Λάιον και να πω ότι εμείς βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της εφαρμογής αυτής της νέας ΚΑΠ. Σήμερα κανένας δεν αμφισβητεί την ανάγκη μιας κοινή αγροτικής πολιτικής, αυτό υπόθηκε. Αλλά θα πρέπει όμως να έχει νομιμότητα αυτή η ΚΑΠ, νομιμότητα έναντι του πολίτη που είναι ο φορολογούμενος είναι αυτοί που χρηματοδοτούν με, τη, με τους φόρους τους στην ΚΑΠ. Πρέπει να υπάρχει λοιπόν μία νομιμότητα για την τροφοδοσία των Ευρωπαίων. Νομιμότητα για την απασχόληση στη Γεωργία. Η γεωργική εκμετάλλευση σήμερα και οι αγρότες σήμερα είναι 12 εκατομμύρια 600 τόσες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Και άμα βάλουμε και τη μεταπητική βιομηχανία είναι άλλα 5 εκατομμύρια ε, θέσεις εργασίας. Παίζουν σημαντικότατο ρόλο λοιπόν στην επικράτειά μας. Χρειάζεται νομιμότητα και για τα θέματα περιβάλλοντος και για τα θέματα ποιότητας. Αυτά πρέπει να τα διασφαλίσουμε, αλλά αν θέλουμε και μία πραγματική νομιμότητα της ΠΑΚ, θα πρέπει, και το λέω στην Κομισιόν, να έχουμε διαφάνεια, συνολική διαφάνεια σε αυτή την ΚΑΠ. Ήδη εμείς συζητήσαμε το θέμα της ε, τροφιμικής αλυσίδας, είναι αυτό που ξεκινήσαμε χθες. Πώς μπορούμε εμεί σήμερα από 31% να έχουμε περάσει στο 21% το μερίδιο των ε, αγροτών ε, στην, των γεωργών στην τροφιμική αλυσίδα για τις τιμές. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σήμερα στις τιμές. Θα πρέπει η Κομισιόν για να μπορέσουμε να δουλέψουμε να απαντήσει στο θέμα της διαφάνειας των τιμών. Σε τρίτο επίπεδο είναι η κατανομή των ενισχύσεων. Πολλοί αναφέρθηκαν στην ανισότητα της κατανομής ε, της ε, βοήθειας μεταξύ αγροτών και κρατών. Μιλάμε σήμερα για πρώτο και δεύτερο πυλώνα, αλλά κανένας δεν μιλάει για το πώς στην πραγματικότητα αυτές οι ενισχύσεις δεν ανταποκρίνονται στους πυλώνες, αλλά ε, στις ε, διάφορες, ε, στα διάφορα κουτιά της ΠΟΕ. Το πορτοκαλί, το πράσινο κλπ. Αν εμεί σήμερα πούμε ότι σταματούμε την επιδότηση των εξαγωγών, η πραγματικότητα θα είναι άλλη, διότι ορισμένες επιδοτήσεις θα περάσουν μέσα από, αυτά τα, από το ένα κουτί στο άλλο κουτί. Δηλαδή θα δοθούν άλλου είδους ενισχύσεις που πάλι επιδοτήσεις θα είναι για τα δημητριακά, για το 8% και κάτι ε, που εξήχθη το 2006 που είναι η τελευταία χρονιά κοινοποίηση στην ΠΟΕ για τις εξαγωγές οι πραγματικές εξαγωγές ήταν ναι, μόνο το 10% των επιδοτήσεων ε, στις εκμεταλλεύσεις. Σήμερα με τα ποσά που δίνονται στην ΠΟΕ οι επιδοτήσεις για τα δημητριακά οδηγούν σε ένα ντάμπινγκ του 61% δεν θα μπορέσουμε εμείς να νομιμοποιήσουμε την πάξη αυτού του είδους την κατάσταση. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και δεν το είπαμε ακόμα τις νέες προκλήσεις που είναι το κλίμα, το νερό και η βιοπικιλότητα. Είναι η χρονιά της βιοπικιλότητας. Θα πρέπει η Κομισιόν να μας δώσει τα νούμερα για τις απώλειες της βιοπικιλότητας που συνδέονται με ένα γεωργικό μοντέλο ανάπτυξης που κατέστρεψε και το έδαφος ε, και το νερό και το τοπίο και όλα. Λοιπόν, πότε θα αρχίσει πραγματικά τη δουλειά η Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο θέλει να δουλέψει, αλλά αυτό θα το κάνει μόνο όταν θα έχει συγκεκριμένα στοιχεία που θα τις δώσει η Κομισιόν. Ευχαριστώ Ζωζέ, πάμε στο δεύτερο πάνελ και δίνω το λόγο στον Αρλίντο Κούνα, πρώην βουλευτή. Ευρωβουλευτή. Σήμερα εμπειρογνώμων στον ακαδημαϊκό πλέον τομέα που μπορεί να μας δώσει τις απαντήσεις. Αρλίντο, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, που με καλέσατε και να ε, χαιρετήσω όλους ε, τους, ε, όλα τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας, πρώην συνάδελφοι και σύντροφοι. Θα ξεκινήσω με βάση πέντε σημεία. Είναι πολύ ευρύ το θέμα, βεβαίω, και δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μα. Αλλά θα αναφερθώ σε, αυτά τα πέντε βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, μπορούμε να αναρωθούμε για το κατά πόσο χρειαζόμαστε ένα ισχυρό και αηφόρο και βιώσιμο γεωργικό τομέα. Ε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στην απάντηση. Η απάντηση είναι καταφατική. γιατί ε, πώς, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, την ε, ασφάλεια στον τομέα της διατροφής, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τις, ε, την προσφορά στην αγορά. Εδώ αναφέρθηκε επίσης το ζήτημα της προστασίας του βιοκυπικιλότητας. Αλλά πρέπει ταυτόχρονα να τονίσουμε τη σημασία της γεωργίας για την οικονομική ανάπτυξη, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Ένα στοιχείο το οποίο το λησμονάμε μερικές φορές. Ε, ε συμβάλλει δηλαδή η γεωργία στην οικονομική και κοινωνική συνοχή. Θέλουμε, δηλαδή, συμφωνούμε ότι θέλουμε ένα ισχυρό ε, γεωργικό τομέα στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Δεύτερο, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε στην Ευρώπη ε, ένα ισχυρό και βιώσιμο γεωργικό τομέα. Πρώτα απ' όλα, αυτό θα το πράξουμε μέσω της ε, ε πολιτικής υπέρ της ανταγωνιστικότητας, μέσω των τιμών, της ποιότητας, της διαφοροποίησης των προϊόντων και ε, αναφέροντας κάθε φορά ε, την προστιθέμενη αξία των προϊόντων αυτών και των, ε, της μεταποίησής τους. Ε, Βεβαίω αρκούσε η πολιτική ε, η δράση προ την κατεύθυνση του ανταγωνισμού, αν είχαμε ένα δίκαιο κόσμο, όπου όλοι ακολουθούσαν του ίδιου κανόνε και όπου δεν υπήρχε αυτή η τεράστια διαφορά σε επίπεδο και αμοιβών. Αλλά δυστυχώ δεν, σε δεν ζούμε σε αυτόν τον ε, ιδεώδη κόσμο. Γι' αυτό η ανταγωνιστικότητα είναι μεν μια απαραίτητη προπόθεση, αλλά δεν είναι η μοναδική προπόθεση. Απαιτούνται και άλλα στοιχεία. Θέλουμε μια δημόσια πολιτική που να εγγυάται ε, ένα σύνολο αγαθών και υπηρεσιών. Τρίτο στοιχείο. με ποιο τρόπο θα, ε, και με ποια επιχειρήματα θα δικαιολογήσουμε την ανάγκη για μια συνεκτική κοινή αγροτική πολιτική ε, στα πλαίσια των αρχών που μόλις ανακοίνωσα. Δηλαδή, ποια θα, είναι η βάση, η ορθολογική βάση του μοντέλου προς το οποίο προσδοκάμε. Ποια θα είναι τα επιχειρήματα που θα συνηγορούν υπέρ του μοντέλου αυτού. Από τη μια λοιπόν θέλουμε μια πολιτική ε, διαρθρωτικής προσαρμογής για να μπορέσει να υπάρξει δυνατότητα προσαρμογής της κοινή αγροτικής πολιτικής στην, ε, στις οικονομικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, και εξωτερικό επίπεδο και για να επιταχυνθεί και η διαρθρωτική προσαρμογή. Αυτό είναι κλειδί για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Γεωργίας. Επίσης ε, χρειαζόμαστε ταυτόχρονα και μια πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική για να, για να προωθήσουμε την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών ε, που δεν αποτελούν αντικείμενο αμοιβή στην αγορά. Δηλαδή, που εμεί θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα, αλλά που δεν ε, ε, τα ανταμείβει επαρκώ η αγορά. Σημαντικό και αυτό. Άλλο θέμα σημαντικό είναι η σταθερότητα σε επίπεδο προσφοράς και εφοδιασμού των αγορών αυτών. Εδώ μιλώ δηλαδή για τη διόρθωση των προβλημάτων των αγορών και των ελλείψεων των αγορών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια δημόσια πολιτική στην Ευρώπη για όλου αυτού του λόγου αν δεν μπορέσουμε ε, να στηρίξουμε την, την κοινή αγροτική πολιτική στα επιχειρήματα αυτά, τότε θα χάσουμε την ευκαιρία και δεν θα μπορέσουμε να ε, αξιοποιήσουμε τα ενδογενή πλεονεκτήματα τα οποία μα προσφέρει η Γεωργία. Θα χάσουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση σε ολόκληρη την επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα προωθήσουμε αντίθετα την ε, έξοδο από την Ήπεθρο την εσωτερική μετανάστευση δηλαδή των ανθρώπων από την Ήπεθρο προς τις αστικές περιοχές. Αυτή που, ε, που πιστεύουν ότι μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα από τον προπολογισμό τη Γεωργία, τελικά τα χρήματα αυτά θα τα χρησιμοποιήσουν για να αντιμετωπίσουν τη μαζική έξοδο από την ύπεθρο και την απερίμωση τη ύπεθρου. Αυτά είναι σημαντικά επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ μια δημόσια και ε, ισχυρή κοινή αγροτική πολιτική. Επόμενη ερώτηση. Ε, η σημερινή κοινή αγροτική πολιτική απαντά με σωστό τρόπο στα ε, προβλήματα τη γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει απαντήσει στα ερωτήματα και στι ανησυχίε των πολιτών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 ανησυχίε κοινωνική φύσεω. Λοιπόν, αν είμαστε ειλικρινεί, θα απαντούσαμε όχι. Η, η σημερινή κοινή αγροτική πολιτική δεν καλύπτει αυτέ τι ε, προσδοκίε. Ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η εξέλιξη τη κοινή αγροτική πολιτική. Πρέπει να πούμε βεβαίω ότι ε, ήταν αφιλεγόμενη, δεν ήταν όλα ρόδινα, αλλά μπορούμε να πούμε ότι η, η πλειοψηφία ε, των ανθρώπων πιστεύει ότι ήταν απαραίτητε αυτέ οι αλλαγέ για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε την κοινή αγροτική πολιτική ε, στη σημερινή κατάσταση. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια ενδογενής έλλειψη στην ΚΑΠ, αυτό που ονομάζω εγώ σχιζοφρένεια. Έχουμε δύο ΚΑΠ. Έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική των πολιτικών και των επαγγελματιών και την άλλη ΚΑΠ, την άλλη κοινή αγροτική πολιτική που είναι ε, η ΚΑΠ ε, επιτόπου, αν θέλετε. Και επιτόπου, αυτό το οποίο αποτελεί αντικείμενο εφαρμογή στα πλαίσια της κοινή αγροτική πολιτική είναι αυτό το, το καθεστώ τη πληρωμής που ακολουθεί ε, τη φιλοσοφία ε, της αποζημίωσης προς τους ε, αγρότες για την πολιτική τιμών που εφαρμόζουμε εδώ και 18 χρόνια. Γι' αυτό με μια κάποια ηρωνία λέω ότι ε, ε, οι είναι η ίδια αλλά η μουσική είναι διαφορετική. Γι' αυτό ε, σας λέω ότι ε, τους, τους αποζημιώνουμε διο, λόγω ακριβώς της μείωσης των τιμών. Και αυτό είναι ουσιώδης σημασία. Αν θέλουμε να εξηγήσουμε στους ε, πολίτες το γιατί η ΚΑΠ δεν ανταποκρίνεται σωστά στα προβλήματα ε, τα οποία αντιμετωπίζει η Γεωργία. Η κοινή αγροτική πολιτική είναι μια πολιτική συνοχής. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε ε, ιδιαίτερα ριζοσπαστικοί για να καταλάβουμε κάτι τέτοιο, αρκεί να κοιτάξουμε τα πρόσφατα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει μια κάποια έλλειψη συνοχής με την ίδια τη συνθήκη. Γιατί ε, πραγματικά έχουμε τη συνθήκη που αναφέρεται ε, στην ε, συνθήκη. Τι θέλουμε λοιπόν σε τελευταία ανάλυση. Θέλουμε μια κοινή αγροτική πολιτική συνεπή με τα ίδια μα τα επιχειρήματα, με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε για να υποστηρίξουμε την ύπαρξή τη, την ανάγκη για την ύπαρξή τη. Και εδώ τώρα, το λέω συχνά αυτό. Πρέπει η θεωρία να συμφωνεί με την πράξη. Αυτό χρειαζόμαστε. Και τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ και σε ένα άλλο θέμα. Τι κοινή αγροτική πολιτική χρειαζόμαστε ε, για το χρονικό διάστημα μετά το 2013, όταν δηλαδή θα έχει ολοκληρωθεί ε, η σημερινή περίοδος που καλύπτεται από τις υφιστάμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Εδώ θέλω να σας πω το εξή. Και ήδη ε, μπήκαμε στην ουσία του ζητήματος. Να σα υπενθυμίσω ότι όσον αφορά τα δημόσια αγαθά, ε, το θέμα αυτό, για το θέμα αυτό θέλω να πω το εξή. Ίσως αν θέλετε το μόνο επιχείρημα το οποίο συνηγορεί υπέρ τη ύπαρξη κοινή αγροτική πολιτική έχει να κάνει με αυτό, με την παραγωγή των δημοσίων αγαθών που ε, παράγονται από κοινού με τα αγαθά τα οποία αποτελούν αντικείμενο εμπορία. Ε, σε μεγάλο μέρος και όχι απόλυτα ε, δικαιολογείται η γεωργία ακριβώς διότι ε, από τη γεωργία παράγονται προϊόντα τα οποία απολούνται στην αγορά. Δεν είναι μουσείο ο κόσμο τη υπαίθρου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αν είχαμε μόνο μία ΚΑΠ η οποία στηρίζεται στην αποζημίωση ε, των ε, δημοσίων αγαθών, για την παραγωγή δηλαδή δημοσίων αγαθών, θα κάναμε λάθος. Δεν έχουμε τη δυναμική αυτή τη στιγμή ε, έτσι ώστε να ψυχώσουμε τους παραγωγούς να εξακολουθούν να παράγουν. θα του αποζημιώνουμε μόνο και μόνο επειδή φροντίζουν το περιβάλλον και το τοπίο. Αλλά αυτό δεν, ε, δεν θα μας οδηγήσει πουθενά. Επιμένω, ε, το ότι είναι, τα δημόσια αγαθά δεν μπορεί να είναι το μοναδικό επιχείρημα. Για να έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική η οποία να μας οδηγεί σε μια ισχυρή και βιώσιμη γεωργία, τότε θα πρέπει να βρούμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα των τιμών και των αποδόσεων. Γιατί ξέρουμε ότι η αγορά είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητη και αυτό χρειαζόμαστε ένα, μια κοινή αγροτική πολιτική που να αποτελεί ένα ελάχιστο δίκτυο ασφαλείας και να βοηθά πραγματικά τους γεωργούς ε, στις περιόδους κρίσης. Εάν δεν έχουμε αυτά τα μέσα στη διάθεσή μας ε, και αν δεν τα δώσουμε προς τον γεωργό ως επιχειρηματία, τότε ο γεωργός δεν θα συνεχίσει τις δραστηριότητε του. Εάν δεν ακολουθήσουμε αυτή την οδό λοιπόν, θα έχουμε βεβαίω μέσα παρέμβαση, τα ίδια, τα παλιά ε, μέσα παρέμβαση και τελικά δεν θα εξυγχρονίσουμε ε, τη δράση μα. Ταυτόχρονα όμω χρειαζόμαστε μια κοινωνικο-διαθετική πολιτική πολύ σημαντική, έτσι ώστε η πολιτική μα να εξακολουθήσει να είναι ανταγωνιστική και ταυτόχρονα χρειαζόμαστε μέσα για να διορθώσουμε τι ε, ε ελλείψει στην αγορά. Τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο. Τελευταίο σημείο τώρα. ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να δούμε όταν μιλάμε για την ΚΑΠ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κοινή αγροτική πολιτική θα πρέπει να έχει στη διάθεσή τη ένα σύνολο ε, μέσων που να χαρακτηρίζεται από ισορροπία και πολιτικών στα πλαίσια τη συνοχή για να μπορέσει να εκπληρώσει του στόχου τη. Η διόρθωση των ε, ελλείψεων των αγορών ε, όταν μιλάμε για δημόσια αγαθά, είναι θέμα το οποίο επίση θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητέ, θα πρέπει να μιλήσουμε για κάποιες ελάχιστες πληρωμές, έτσι, για να ε, υπάρξει αποζημίωση για διαφορές που υπάρχουν άμεσα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις τρίτες χώρες, εκεί όπου οι κανόνες δεν είναι τόσο πολύ αυστηροί όσο στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πρώτο επίπεδο που είναι ε, η, η πολλαπλή συμμόρφωση και στη συνέχεια έχουμε και ένα δεύτερο επίπεδο που αφορά την ε, πληρωμή αυτή για τα εξαιρετική σημασία δημόσια αγαθά. Και αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο το επίπεδο πληρωμών θα πρέπει να είναι το ίδιο σε, όλο, σε όλη την επικράτηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ξέρετε, ε, το επίπεδο αυτό ε, ενίσχυση προ του γεωργού διαφοροποιείται. Βεβαίω, το ιδεώδε θα ήταν να ήταν το ίδιο, αλλά γνωρίζουμε ότι η μισθή και το βιωτικό επίπεδο σε διάφορε χώρε μέλη δεν είναι το ίδιο. Γι' αυτό ε, οι, οι, οι πληρωμέ αυτέ θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τι διαφορέ του βιωτικού επίπεδου, παρόλο που θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση αυτών των επιπέδων. Θέλουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο σύγκληση, το οποίο αποκτά όλο και περισσότερη σημασία. Αυτό όμω το οποίο δεν είναι καθόλου πιθανό είναι να εξακολουθήσουμε ε, να μεγεθύνουμε τι ανισότητε ανάμεσα στην αμοιβή των γεωργών στην Α χώρα και στη Β χώρα. Μερικέ φορέ οι διαφορέ ε, είναι από το 1 ω το 20, αν θέλετε. Πρέπει λοιπόν να διορθώσουμε μία σειρά από ελλείψεις γιατί μια πιο ισότιμη κατανομή ε, των ενισχύσεων τη κίνηση αγροτική πολιτική αποτελεί απαραίτητη προπόθεση για να καλυφθούν οι ε, ανισότητε και οι ελλείψη αγορά. Εάν δεν πετύχουμε αυτή την, τη μεγαλύτερη δικαιοσύνη στον επιμερισμό των ενισχύσεων στου γεωργού, τότε σα το λέω από τώρα, δεν θα μπορέσουμε να ε, υπερασπίσουμε την ύπαρξη μια πολύ πιο ισχυρή γεωργία. Διότι στην αντίθετη περίπτωση όλα τα επιχειρήματα υπέρ μια ισχυρότερης γεωργίας θα ε, είναι απλή ρητορική και τίποτα περισσότερο. Και το μόνο προχωρήσουμε, να προχωρήσουμε και περισσότερο. Η προάσπιση τη κοινή αγροτική πολιτική έναντι των πολιτών και τη κοινωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να, γίνει, ε, να είναι εφικτή αν δεν ζητήσουμε περισσότερη δικαιοσύνη τη στιγμή τη κατανομή των ενισχύσεων στου γεωργού. Γιατί αυτέ οι διαφορέ, καταλαβαίνετε, ότι θα, θα στρεβλώσουν το μήνυμα που θέλουμε να εκπέμψουμε προ Ευρωπαίου πολίτε. Και οι Ευρωπαίοι πολίτε θα καταλαβαίνουν όλο και λιγότερο γιατί πρέπει να πληρώνουν την κοινή αγροτική πολιτική. Και επειδή προφανώ όλο και περισσότερο θα υπάρχουν περισσότεροι τομεί και περισσότεροι ανταγωνιστέ ε, που θα θέλουν ε, να ε, πάρουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο του προπολογισμού, η θέση των γεωργών θα επιδεινώνεται όλο και περισσότερο. Τελειώνω λέγοντά σα ότι η ενίσχυση με βάση τα εκτάρια δεν αντικατοπτρίζουν ε, τα, αυτό το γεγονό ότι πρόκειται για δημόσια αγαθά, τα αγαθά που παράγονται από τη Γεωργία και θα πρέπει να μην ακολουθήσουμε αυτά τα κριτήρια, αλλά άλλα, κοινωνική φύσεω, περιβαλλοντική φύσεω ή ε, κριτήριο πρόθεση απασχόληση. Και επίση αναφέρθηκε εδώ και το θέμα τη ε, ε, ε χρηματοδοτική αλληλεγγύη, δηλαδή η συγχρηματοδότηση ε, κοινοτική. Και να σα πω το εξή σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Για μένα το σημαντικό δεν είναι σημαντικό το αν ε, η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου τη ΚΑΠ προέρχεται, οφείλεται μάλλον στον πρώτο πυλώνα ή στο δεύτερο. Το σημαντικό είναι να επιτευχθεί ο στόχο. Αν εγώ πληρώνω για την παραγωγή ενό ε, δημόσιου αγαθού, δεν με ενδιαφέρει το κατά πόσο αυτό γίνεται στα πλαίσια του πρώτου του δεύτερου πυλώνα. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ο συγκεκριμένο στόχο. Και μάλιστα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η διαφορά ανάμεσα στον πρώτο πυλώνα και στο δεύτερο πυλώνα σιγά σιγά θα αρχίσει να εξαλείφεται και στο δεύτερο πυλώνα στη συνέχεια θα μείνει αυτό το οποίο ονομάζουμε ανάπτυξη πέθρου. Τελικό συμπέρασμα μακροπρόθεσμα μπορούμε να υπερασπίσουμε την ΚΑΠ μόνο αν είναι μια συνεκτική πολιτική. Πράγμα που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια συνεκτική πολιτική. Και αν θέλουμε να την αλλάξουμε, να την αλλάξουμε. Αλλά ε, στα πλαίσια αυτά της υποστήριξης. αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κούνια. Συνεχίζουμε με τον κύριο Λουί Πασκάλ Μαέ, καθηγητή στο... στη Ρένα, στο Πανεπιστήμιο, στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο της Ρένα, για να μας μιλήσει για ένα νέο πρότυπο για τη Γεωργία. Έχετε το λόγο κύριε Μαέ. Merci, Monsieur le Président. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η παρουσίασή μου αφορά σε ένα νέο σύστημα πληρωμών για την ΚΑΠ για μετά το 2013. Η παρουσίαση βασίζεται σε προηγούμενες εργασίες και τις που το έχετε και στο έγγραφό σας των 7 σελίδων που λάβατε προηγουμένως. Να σας τα αναφέρω όμως, είναι ουσιαστικότατα αυτά. Είναι η έκθεση για την Ένωση Notre Europe ε, του Jacques Delors με συνεργάτη τον κύριο Μπυρό και που λέει τα ίδια πράγματα που είπαμε χθες. Λοιπόν, μερικές σύντομες παρατηρήσεις τώρα για τα, ε, για τα καλά αλλά και για τα όρια τα οποία έχει η ΚΑΠ. Να σας αναφέρω επίσης το τι βλέπουμε για το 2013 αλλά θα αναφερθώ μόνο στη διάρθρωση των ε, άμεσων πληρωμών Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζονται θεσμοί για να αντιμετωπιστεί η αστάθεια των τιμών και των εισοδημάτων. Εγώ θα ήθελα να έχουμε και ένα δίχτυ ασφάλειας για τις τιμές με όρους που δεν έχω το χρόνο να σας αναπτύξω. Και απ' την άλλη το έπανε και άλλοι ομιλητές και το προσυπογράφω, χρειάζεται να έχουμε θεσμούς για να ενισχύσουν της, ε, το μερίδιο αγοράς των αγροτών που είναι πολύ αδύναμο διαφορετικά. Υπάρχουν ε, βέβαια πράγματα που στην κοινή οργάνωση των αγορών, στις ΚΟΕΣ, που θα πρέπει να τα διατηρήσουμε, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ της δεσπόσας θέσης των ολιγοπολίων και των οργανώσεων των αγροτών. Οι προηγούμενες ε, μεταρρυθμίσεις ήταν ε, κυρίως αλλαγές μέσων που διόρθωναν τις, ανισορροπ... τις ανισορροπίες των βασικών εσωτερικών αγορών και που μείωσαν εν μέρη την εντατικότητα της γεωργίας. Αλλά αυτές οι αλλαγές ήταν ε, σχετικά περιορισμένες και ως προς το επίπεδο και ως προς τον τρόπο κατανομής της υποστήριξης μεταξύ των γεωργών. Το μέγεθος της εκμετάλλευσης στο γεωργικό σύστημα μετράνε πολύ περισσότερο από τις γεωργικές πρακτικές, που σήμερα όμως είναι πολύ σημαντική πρόκληση. Κατά συνέπεια η ποιότητα του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη της υπαίθρου είναι δύο προκλήσεις που δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά. Είναι αμφίσιμα τα, περιβαλλοντικά ευεργετήματα των μεταρρυθμίσεων. Ο απολογισμός δε των ε, σχεδίων ανάπτυξης της υπαίθρου και η επίδρασή του στην απασχόληση είναι επίσης ε, αρκετά χαλαρά ε, ε, εκεί όπου εφαρμόστηκε αυτή η πολιτική, ίσως εκτός από τις ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Οι βελτιώσεις όμως δεν αλλάζουν ε, τη λογική των άμεσων πληρωμών, κυρίως με την ενιαία εισφορά Έχουμε λοιπόν τα διάφορα δικαιώματα που δίνουν πρόσβαση στην ενίσχυση, τα οποία δικαιώματα είτε χορηγούνται από το κράτος, είτε είναι κληρονομικά και δεν δίνονται βάση των προσδοκιών της κοινωνίας και δεν επίσης ε, ξεφεύγουν από το προπατορικό αμάρτημα που είναι η λογική της αντιστάθμισης. Και επίσης δεν είναι και πολύ θέλκτη και τα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος τα οποία δεν έχουν καμία συνάφεια, είναι εντελώς άσχετα με τους ε, στόχους που έχουμε. Τώρα για την αποτελεσματικότητα στην πράξη της ε, της οικοπολαπλής συμμόρφωσης Ναι. Διότι μας, βγάζουν, μας, εντάσσουν μια κουλτούρα η οποία δεν είναι απόλυτα σύμβατη με την κατάσταση σήμερα. Επίσης δείχνει και μια πολιτική αδυναμία της Ευρώπης η οποία δεν αντιμετωπίζει ευρωπαϊκά τα δικά της προβλήματα και αυτό είναι θλιβερό. Τελευταίο σημείο. Ο περιορισμός της χρηματοδότησης στα μέτρα του δεύτερου πυλώνα δεν διασφαλίζει σαφώς την ευθύνη των κρατών μελών. Υπάρχουν και διαφωνίες, σημαντικές διαφωνίες στα θέματα του δευτέρου πύλωνα. Παίζεται μια εσωτερική τραγωδία στο πεδίο αυτό. Η αλληλεγγύη, η, η, οικονομική αλληλεγγύη επίσης δεν στέκεται έτσι όπως έχει. Χρειάζεται μια νέα αντίληψη, χρειάζεται ένα νέο ξεκίνημα και η συνθήκη της Ρώμης θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Βέβαια εντάξει χάσαμε την ευκαιρία αλλά στο μέλλον Όμως βέβαια αυτήν την ανάγκη την αναγνώρισε το Συμβούλιο των Υπουργών. Η εισοδηματική υποστήριξη παρά την υπάρχουσα κρίση δεν είναι επαρκές επιχείρημα για την άμεση ενίσχυση. Σίγουρα η οικονομική σιγουριά είναι κάτι το, το, που στέκει ως ε, επιχείρημα. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί και να αξιοποιήσουμε πραγματικά τα μέσα που έχουμε, δεν στέκει μόνο του αυτό το επιχείρημα. Δεν θα πρέπει εμείς να μπερδεύουμε τη σταθεροποίηση με τα πρακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Δεν μπορούμε εμείς να συνδέουμε μακροπρόθεσμα την άμεση ενίσχυση με την τωρινή κρίση, την κυριακή κρίση. Θα πρέπει να δούμε πού είναι τα προβλήματα της τωρινής, των τωρινών αγορών. Το δημόσιο χρήμα θα πρέπει να τεθεί σε υπηρεσίες που αφορούν στην κοινή ωφέλεια, περιβάλλον κλπ. Θα πρέπει τα δημόσια χρήματα να αμείβουν δημόσιες πρακτικές. Προτείνω λοιπόν κατά συνέπεια τα εξής. Διαφοροποίηση, στόχος, αναλογικότητα, αποτελεσματικότητα, συνάφεια. Ας πούμε θα πρέπει να είναι πιο θελκτικές οι ενισχύσεις προς τη βιολογική γεωργία από ό,τι προς τη συμβατική συμβαίνει το αντίθετο σήμερα. Απλούστευση και σταθερότητα, μείωση του διοικητικού κόστους. ελευθερία σύναψη συμβολέου. και όχι ενισχύσεις ανοιχτή θηρίδας. Έχουμε λοιπόν ε, δημόσιο χρήμα το οποίο επίσης θα πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίζουμε και το σεβασμό των ατόμων. Ε, επίσης, ευθύνη, οικονομική ευθύνη των κρατών μελών. Έχουμε δύο λοιπόν βασικές προκλήσεις, καλύτερη διάρθρωση μεταξύ εννέας πληρωμής και κινήτρων για να διατηρήσουμε το δημόσιο αγαθό της υπαίθρου και να πειθαρχήσουμε, να τακτοποιήσουμε τις κρατικές προθέσεις και τις κρυφές σκέψεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Να έχουμε λοιπόν ε, μία βασική πληρωμή η οποία θα έχει ως στόχο τη συμβατική γεωργία προς τις που θα στρέφεται προς τις αγορές σε μπανάλ περιοχές, δηλαδή τις περισσότερες, ε, την περισσότερη επικράτεια Θα έχουμε δηλαδή μειωμένες άμεσες πληρωμές, οι οποίες ούτε θα πουλούνται ούτε θα δίνονται σε κληρονομιά, θα έχουν μια περιορισμένη διάρκεια, αλλά μακρόχρονη περιορισμένη διάρκεια. Είπαμε επίσης αμοιβή των υπηρεσιών του για το κοινοφελές έργο, ανάλογα με τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα επιχείρημα διαφοροποίησης που δεν αντιβαίνει με τη σύγκληση μακροπρόθεσμα. Δεύτερη φάση, οι πληρωμές για φυσικά εμπόδια. Δηλαδή στην Ήπεθρο που έχει προβλήματα φυσικά προβλήματα και που δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική και η οποία όμως είναι απολύτως απαραίτητη για τον ε, οικονομικό ιστό της υπαίθρου. Αυτή η πληρωμή μπορεί να συνδυαστεί με την παραγωγή Βέβαια αυτό το ζευγάρωμα των ε, δύο πριμ δεν, μπορεί, δεν μπόρεσε μέχρι τώρα να λειτουργήσει αλλά θα πρέπει να οριστεί αυστηρά και αυτό λόγω της ουσιαστικής, ε, του ουσιαστικού ρόλου της γεωργίας ε, στην τοπική ανάπτυξη. Σε τρίτη φάση πληρωμές, οι πράσινες πληρωμές που θα πληρώνουν τις επιχειρήσεις, τις εκμεταλλεύσεις εκείνες οι οποίες δεσμεύονται για την παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών. Αυτές οι πληρωμές θα έπρεπε να είναι αντίστοιχες με συσσωρευμένα σημεία, με πόντους που θα μαζεύουν οι επιχειρήσεις, και θα έπρεπε να δίνονται στις περιοχές εκείνες που έχουν ιδιαίτερο ευπαθές περιβάλλον και θα μπορούσαν αυτές οι Αυτές οι εκμεταλλεύσεις σε αυτούς τους υπέ, στις υπαίθριες περιοχές να αμβλύνουν το ρόλο της εντατικής γεωργίας. Δηλαδή, προστασία των υδάτων και ευπαθών περιοχών. Να έχουμε συμβόλαια, όχι κατευθείαν πληρωμή στον ΚΙΣΕ. τα δικαιώματα δεν θα διαβιβάζονται. Και αντί οικονομική ελληνική θα πρέπει να έχουμε μία δεσμευτική αλληλεγγύη. Να έχουμε συγκεκριμένα συμβόλαια. Δέσμευση λοιπόν. που θα περιορίσει την απληστία των κρατών που βλέπουν μέσα από τη χορήγηση του καθαρού υπόλοιπου τρόπο για να μπαλώσουν τα δικά τους ελλείμματα. Συμπέρασμα. Είπαμε πληρωμή συμβολέων με τρόπο ad hoc και ρεαλιστικά. Αυτό δεν θα πρέπει να υποκαταστήσει τις άλλες πολιτικές, περιφερειακή πολιτικές ή πολιτικές ανάπτυξης της υπαίθρου ή προστασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει επίσης να μειωθεί το διοικητικό κόστος. Δηλαδή, το κόστος των, των διοικητικών υπηρεσιών και της υπηρεσίας που παρέχεται είναι δυσανάλογο. Χρειάζεται λοιπόν και αυτό να διορθωθεί και να ληφθούν υπόψη και οι διαφορές μεταξύ των χωρών. Επίσης, χρειάζεται υπερεθνικότητα για την ΚΑΠ διότι τα κοινά αγαθά της υπαίθρου, βιοπικιλότητα, κλίμα, περιβάλλον και όλα αυτά είναι κοινά αγαθά. Και υπάρχει βέβαια και η λογική της επικουρικότητας που παρεμβαίνει, δεδομένου ότι οι παρεμβάσεις γίνονται τοπικά. Και η χρηματοδότηση επίσης χρειάζεται. Ο φορολογικός φεντεραλισμός δεν αυξάνει τις ικανότητες τοπικά ας πούμε το νερό προστατεύεται είναι μια οικονομική αξία, από την άλλη μεριά έχουμε ηθικές αξίες, προστασία της βιοποικιλότητας. Είναι κάτι λοιπόν που θα πρέπει να το δει κανείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όπως τα παρουσιάζαμε κάποτε. Και για να τελειώνω, συμπερασματικά χρειάζεται μια κοινή πολιτική, λιγότερο όμως λερωμένη από τα εθνικά συμφέροντα για τα καθαρά υπόλοιπα. Δεύτερον, η Ευρώπη χρειάζεται τους γεωργούς της, όχι μόνο για την παραγωγή τροφίμων, αλλά για τη διατήρηση του μοντέλου της του μοντέλου της υπαίθρου που είναι μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς. Η συλλογική δράση είναι πολύ καλά οργανωμένη για να προασπιστεί ε, η ευημερία της ε, γεωργικής κοινότητας, αλλά αυτό δεν συμβαίνει για τα υπαίθρια κοινωνικά αγαθά που δεν έχει, ε, για τα οποία δεν υπάρχει εκλογικό σώμα του χρήστη. Χρειάζεται λοιπόν μια καλύτερη κάπα, πιο στοχευμένη ε, για το καλό των γεωργών αλλά και για τους υπόλοιπους και την Ευρώπη γενικότερα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ καθηγητά. Λουί Πασκάλ Μαέ. Τελειώνουμε λοιπόν με τους εμπειρογνώμονες. Ο Αντρέι Κοβάλσκι έχει το λόγο, καθηγητής της Βαρσάου School of Economics στο Ίδρυμα Γεωπονικής. Γιατί η ΚΑΠ θα πρέπει να συνεχίσει να παραμένει ευρωπαϊκή πολιτική, το λόγο καθηγητά Κοβάλσκι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. κύριε και κύριοι. Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε με την πρόσκληση να έρθω σήμερα εδώ στις συζητήσεις. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ως τελευταίος ομιλητής, ύστερα από τόσους μεγάλους ρήτορες που προηγήθηκαν, αισθάνομαι αμηχανία διότι έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα. Πολύ λίγα πράγματα έχω εγώ να προσθέσω. Κύριε Πρόεδρε, ίσως θα μπορούσα να ξεκινήσω με μια προσωπική νότα και ανεκδοτολογικά να σας πω ότι όποτε έχω επισημάνει συζητήσει μου ότι ασχολούμαι με την γεωργική οικονομία, μου λένε όλοι Ξέρεις πώς να χάνεις χρήματα δηλαδή. Εκπλήσουμε λοιπόν και μου λένε να σου εξηγήσω. Τρεις τρόποι να χάσεις χάνεις χρήματα. Να παίζεις στο καζίνο, ο πιο γρήγορος και εγγυημένος τρόπος. Ο δεύτερος ε, πληρώνοντας για σεξ, πράγμα το οποίο προσφέρει όμως και μια σχετική ικανοποίηση. Και τρίτον, γεωργία, ο πιο ασφαλής τρόπος να χάσει χρήματα. Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει ότι ο τρίτο τρόπο δεν οδηγεί σε απώλεια χρημάτων. Έχει αποδειχθεί ότι δεν ευσταθεί αυτή η δήλωση. Η πολιτική για την ύπεθρο στην Ευρώπη, η γεωργική πολιτική στην Ευρώπη πρέπει να παραμείνει κοινή. Αυτό θα προσπαθήσω και εγώ να εξηγήσω για να καταρρύψω το τρίτο σκέλος του ανεκδότου. οι διαφορές ε, απόψεων που διαπιστώνονται μερικές φορές, ε, ε, ίσως οφείλονται στο γεγονός ότι η γεωργική πολιτική προσδιορίστηκε μέσα από τη συνθήκη της Ρώμης, χωρίς όμως μετά να δοθεί ποτέ νέος κοινό ορίσμος αυτής της πολιτικής. Ίσως λοιπόν έχει έρθει η ώρα να συζητήσουμε διεξοδικά τι σημαίνει κοινή γεωργική πολιτική. Και ένα καλό σημείο κίνησης πιστεύω θα ήταν ένας ορισμός που βρήκα σε ένα γαλλικό ε, εγχειρίδιο και ο οποίος έχει ως εξής κοινή ορική πολιτική είναι ένα βασικό θεσμικό πλαίσιο μέτρα και κονδύλια για την υλοποίηση των μέσων αυτών. Και οι κοινές πολιτικές θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια πολιτική και κονδύλια που όμως δεν θα θέτουν ένα αμφιβόλο είτε της, ε, την εθνική ε, συνεισφορά, την εθνική συνιστόσα, είτε την κοινοτική συνιστόσα σε σχέση με τις συναλλαγές με τρίτες χώρες. Ε, σε σχέση λοιπόν με την κοινή γεωρική πολιτική νομίζω μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε ότι σύν χρόνο η πτυχή της, του κοινού, η, έννοια, η λέξη κοινή, ξεχάστηκε κάπου, Λυσμονήθηκε. Ίσως αυτό οφείλεται στην ε, ΓΚΑΤ, στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις εξελίξει εκεί. Περαιτέρω διευρύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης τα συμφέροντα των κρατών μελών και ο ενισχυόμενος διαρκώς ρόλος ε, του δεύτερου πυλώνα και τα μέτρα της ε, διαφοροποίησης οδήγησε σε μια διάβρωση που οδηγούν ορισμένου στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να επανεθνικοποιηθεί η γεωργική μας πολιτική. Αυτό βεβαίως για να το συστήσουμε θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τις παραδόσεις και την ιστορία της Ευρώπης και της Γεωργίας στην Ευρώπη. Δεν μπορεί δηλαδή η ε, ποικιλότητα, η ποικιλομορφία την οποία παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Γεωργία να σημαίνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν κοινοί στόχοι. Οι κοινοί στόχοι θα πρέπει να διεκδικήσουν, να εξασφαλίσουν καλύτερη γεωργία, καλύτερα προϊόντα, καλύτερη ανταγωνιστικότητα. Και ένα από τα παραδείγματα ε, από τις, ε, τα επιχειρήματα καλύτερα υπέρ τη επανεθνικοποίηση είναι το κόστος, Γιατί προβάλλεται το επιχείρημα ότι με την επανεθνικοποίηση μειώνεται το κόστο. Χώρες πλούσιε που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ελβετία, η Νορβηγία, το... η Ιαπωνία, πολλές φορές επισημαίνουν ότι οι δαπάνες γεωργικε ίσως είναι υψηλότερες ε, από αυτές τις οποίες καταγράφουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές η επανεθνικοποίηση της γεωργικής πολιτικής κινδυνεύει να οδηγήσει σε δαπάνε πολύ υψηλότερες από αυτές τις οποίες έχουμε ήδη ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έτσι η επαναθνικοποίηση δεν είναι λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον δε, Δεδομένου ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ή άλλε χώρε, ενώ μα υποδεικνύουν κάποιε πολιτικέ, δεν τι εφαρμόζουν οι ίδιε. Αυτό σημαίνει ότι ε, δεν είναι εφαρμόσιμε προφανώ. Έτσι λοιπόν, το 2007, 12 χώρε παρουσίασαν κόστος παραγωγής υψηλότερο από τις τιμές της αγοράς. παρά την κοινή γεωργική πολιτική. Και μάλιστα δέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο στο μέλλον ο αριθμό τέτοιων ε, χωρών που παρουσιάζουν τέτοιε επιδόσει. Βέβαια, η διατήρηση τη κοινή γεωργική πολιτική στην Ευρώπη δεν σημαίνει ότι μπορεί αυτή η πολιτική ή ότι θα πρέπει να παραμείνει απαράλλακτη. Όχι, του αντίδειον, όχι μόνο μπορεί να αλλάξει, αλλά πρέπει και να αλλάξει για να ανταποκριθεί σε νέες προκλήσεις. Υπάρχουν διάφορες πτυχές που χρειάζονται περαιτέρω εναρμόνιση τόσο ως προς τις εθνικές πολιτικές αλλά και ως προς τις ε, ευρωπαϊκές. Καταρχάς θα πρέπει να διαφυλαχθεί το δυναμικό της γεωργικής παραγωγής προκειμένου να εξασφαλιστεί να διαφυλαχθεί η ε, πιστιστική ασφάλεια στην Ευρώπη αλλά και να ικανοποιηθούν οι αυξανόμενες ολόκληρο τον κόσμο επιστηστικές ανάγκες. Η Κατά την άποψή μου όμως δεν μπορεί να διατηρήσει, να εξασφαλίσει μάλλον την ανταγωνιστικότητα για την ιστορική αγορά. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος, άλλο ένα σύστημα με τη διαχείριση των αγορών και τον περιορισμό των σημαντικών κοιμάνσεων των αγορών ε, στην, ε, στα γεωργικά προϊόντα που θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω πιστεύω. Και επίσης θα ήταν χρήσιμο να εξεταστεί και να προωθηθεί η απλούστευση των όρων εφαρμογής των διατάξεων της ΚΑΠ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε με προκλήσεις. Τις λησμονούμε μερικές φορές και ε, κοιτάμε μόνο, στρεφόμαστε το βλέμμα μόνο στα νέα κέντρα κατανάλωσης. Ωστόσο, υπάρχουν και νέα κέντρα κατανάλωσης Γιατί μην ξεχνάτε παραδείγμα ότι πριν από 20 χρόνια κανείς δεν θεωρούσε την Κίνα ως ένα σοβαρό νέο κέντρο κατανάλωσης. Πού έχουμε φτάσει όμως τώρα, πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αναπτύσσονται διαρκώς νέες τεχνολογίες, αναπτύσσονται τα λεγόμενα εφή τρόφιμα σε ολόκληρο τον κόσμο και η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Τώρα δεν θα επεκταθώ σε πράγματα τα οποία ήδη εξετάθησαν ε, από του προηγούμενου ομιλητέ. Θα ήθελα απλώ να υπογραμμίσω ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιδράσει και στι οικολογικέ προκλήσει, προκλήσει του μέλλοντο. Και είμαι πεπισμένο ότι ακόμη και η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης μόνη της δεν θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις. Κυρίες και κύριοι, ως εκπρόσωπος νέου κράτους μέλους θα ήθελα να πω μερικά λόγια για την κοινή πολιτική και την προοπτική ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη. Απευθύνομαι προκειμένου στους περισσότερους ε, ε, εκπροσώπους των παλαιότερων κρατών μελών. Ξέρετε λοιπόν πόσο ακριβή είναι η γεωργία. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για χώρες με πολύ χαμηλότερο ΑΕΠ από τις πλούσιες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρήσουν κάποια καλά επίπεδα στην παραγωγή τους. Και πέραν αυτού τα νέα κράτη-μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν και την εσωτερική ε, τον ιστορικό ανταγωνισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχρεωμένα δηλαδή να τηρήσουν τη στρατηγική της Λισαβόνας. Μερικές φορές προβάλλεται το επιχείρημα αυτό και στι στις πολιτικές συζητήσεις. Έχει έρθει όμως πλέον η στιγμή να θέσουμε ένα τέλο στην ε, αναδιάρθρωση της ε, πρέπει να αναπτύξουμε τι νέε τεχνολογίε κτλ. Αυτό είναι διάφορα επιχειρήματα που ακούγονται, αλλά θέλω, θέλω να πω εγώ ότι εάν από, με, από όλη αυτή την προσπάθεια το αποτέλεσμα που θα βγει θα είναι η ε, απώλεια της κοινή διάστασης για την ε, γεωργική πολιτική, ίσως όχι η Πολωνία η οποία δεν έχει τόσο πολύ πληγή από την ε, οικονομία, την οικονομική κρίση, αλλά άλλες χώρες οι οποίες έχουν ε, υποστεί σημαντική σημαντικό περιορισμό ω προς, ε, προς το ΑΕΠ του. έχουν χάσει ε, αρκετές μονάδες από το ΑΕΠ του. κινδυνεύουν να μην έχουν επαρκή μέσα για να χρηματοδοτήσουν ε, την πολιτική του στη γεωργική, μεταξύ άλλων. Άλλωστε έχουμε δει και πως συνεδριάσει με ε, γεωργούς, όπως συζητούμε τις προκλήσεις, ότι μας λένε πως 40 με 50% σε σχέση με την ε, ε, προενταξιακή περίοδο ήταν η απώλεια εισοδήματος. Και καταλήγω με ένα σχόλιο ότι μερικές φορές τα κράτη-μέλη ε, τα νέα κράτη-μέλη καλύτερα αντιμετωπίζονται σαν τα κράτη-μέλη τα οποία δεν κάνουν αρκετέ προσπάθειε, δεν έχουν προχωρήσει επαρκώ τι μεταρρυθμίσει του. Όχι, εγώ θα σα πω ότι η Πολωνία έχει ξεκινήσει με ένα πληθωρισμό τη τάξη του 2.000% πριν να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο ω χώρα να ανησυχούμε μην πάει στο 4% προπολογισμό ο πληθωρισμό μα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, τι μεγάλη πρόοδο έχουμε κάνει, αλλά φανταστείτε τι σημαντικό κοινωνικό κόστος είχε όλο αυτό. Και επίσης, φανταστείτε ότι χρειάστηκε να δεχθούμε και μεγάλες αλλαγές στην κοινωνική πολιτική και όχι αυτά που θα θέλαμε τέλο πάντων ως προς τη γεωργική μας πολιτική. Αναγκαστήκαμε να δεχθούμε όλα, ε, όλους αυτούς τους δυσμενείς όρους έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά, από το δικό μας μετερίζει, την κοινή γεωρική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ καθηγητά Κοβάλσκι για την παρουσίαση. Τελειώσαμε με την ακρόαση. Η κυρία Κλάσσα έχει το λόγο για το δεύτερο τμήμα της συζήτησης. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμε Πρόεδρε κυρίες και κύριοι. Είδαμε πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρουσιάσεις, ε, συζητήσεις ε, εκπροσώπους της γεωργικής πολιτικής και από το χώρο της γεωργίας και από το χώρο της οικονομίας υπόθηκε από τον κύριο Κούνιο ότι πρέπει να, κάνουμε, πρέπει να είμαστε θέση να παράγουμε τα προϊόντα αυτά τα οποία χρειάζεται η κοινωνία μας. Είμαι βέβαιη και εγώ ότι είμαστε σε θέση να παραγάγουμε να παράγουμε τα προϊόντα που χρειαζόμαστε, τα καλά προϊόντα που χρειάζεται ο πολίτης, αλλά ταυτόχρονα να διαφυλάσσουμε και το ευρωπαϊκό τοπίο, την ευρωπαϊκή ε, ύπεθρο. Άρα παράγοντας με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ήδη μία προσθέμενη αξία. Αυτό θα έπρεπε να ισχύει, ωστόσο υπόθηκε ήδη ότι οι ε, σημαντικές πιέσεις από τις κλιματικές αλλαγές ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό της κοινής γεωργικής πολιτικής. Επίσης, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι η γεωργική πολιτική γεωργία θα πρέπει και αυτή να υποστεί τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Εδώ θα ήθελα να πω εγώ ως ευρωβουλευτή ότι στην Επιτροπή Περιβάλλοντος θέσαμε τα ερωτηματικά αυτά στην Επιτρόπο Χίντεγκάρτ η οποία πολλές φορές πρέπει να σημειώσω επανειλημμένως είπε ότι συμβάλλει και πρέπει να συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία η γεωργία και μάλιστα επισήμανε κάποιες πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Δανία ε, που επιτρέπουν συστηματικά να ε, συμπεριλαμβάνεται η κλιματολογική διάσταση, η περιβαλλοντική η κλιματολογική διάσταση στην γεωργική πολιτική. Στη Δανία τουλάχιστον η κυρία Χιντρίκαρτ μας είπε ότι θέλει μια πράσινη γεωργία. Την, ε, παραθέτω εδώ τα λόγια της, είπε ότι μια τέτοια πράσινη γεωργία μπορεί να είναι και ουδέτερη οικονομικά αυτό νομίζω ότι είναι μια πρόκληση για τους οικονομολόγους εδώ, κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν κάποια σημεία εκκίνησης, κάποιες βασικές ιδέες που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε περισσότερο. Και επίσης θα ήθελα να γνωρίζω και αν γεωργοί πιστεύουν ότι μπορούμε να έχουμε μια ε, δίκαιη κατανομής των απολογισμών για το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτές λοιπόν τις ανησυχίες θα πρέπει να τις συμπεριλάβουμε στη συζήτηση. Θα ήθελα με την ευκαιρία να, τους, να ακούσω τις απόψεις των ειδικών σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα συνεχίζουμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Να ζητήσω από όλου του συναδέλφου που θέλουν να πάρουν το λόγο να είναι πάρα πολύ σύντομοι. Δύο λεπτά το πολύ ο καθένα, γιατί έχω ένα μακροσκελέστατο κατάλογο. Κυρία Μαγκίνε έχει το λόγο. Thank you. I hope... Ευχαριστώ. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε ε, οι παρατηρήσει σα ε, να μην αφορούσαν εμένα προσωπικά. Πάντω προσπαθήσω και να είμαι σύντομη. Δεδομένη τη δήλωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συνολική κατάρρευση του εισοδήματο των γεωργών και παραθέτω τα τελευταία δύο χρόνια, 2008 και 2009, η απώλεια εισοδήματο ήταν τέτοιε. Ε, με άλλα λόγια, δηλαδή δεν θα έχουμε τα, ε, ε, τα, τα, τα, εισοδήματα τα οποία είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση, δηλαδή, από άποψη εισοδηματική. Και ω απορία θα ήθελα να κάνω τι εξή παρατηρήσει κάποιο, στην Επιτροπή μας ιδιαίτερα, θα πρέπει να μην ακολουθήσει τον αποδεκτό κανόνα ότι ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται απειλή και ότι πρέπει να δεχτούμε περικοπέ. Δεν πρέπει να δεχτούμε περικοπέ του γεωργικού προπολογισμού. Και δεδομένη πραγματικότητα των εισοδημάτων των γεωργών, που μόλι ε, τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να ζητήσουμε αύξηση του γεωργικού προπολογισμού. Σα παρακαλώ, ε, μην ε, αρχίζουμε τώρα να χρησιμοποιούμε πρόσχημα τον προπολογισμό. Δεύτερο, α σταματήσουμε να κάνουμε συγγνώμη για την κοινή αγροτική πολιτική. Α σταματήσουμε να ακούμε αυτού που λένε πρέπει να πείσουμε το κοινό για την κοινή αγροτική πολιτική. Μα οι πολίτε υποστηρίζουν τη γεωργία ε, και ε, ε, με, με τι δικέ του αγορέ έχουν, πάρει τι αποφάσει του όσον αφορά τι τιμέ που θα πρέπει να δώσουν για τα δημόσια αγαθά και τα υπόλοιπα και μέσα του συστήματο τη φορολογία. Αυτά είναι δεδομένα. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε σκληρότεροι στον τρόπο με τον οποίο αγωνιζόμαστε. Και να ε, υποστηρίξουμε ε, και τους γεωργούς και την ε, βιομηχανία των τροφίμων. Χθε συζητήσαμε το θέμα, συνολικά το θέμα των δημοσίων αγαθών. Και ειλικρινά δεν μπορώ να δεχθώ ότι αυτή τη στιγμή ζητάμε από του γεωργού να κάνουν περισσότερα για λιγότερα χρήματα. Δεν είμαι σίγουρη όμω για το οποίο δέχομαι ταυτόχρονα απόλυτα την έννοια ότι δεν μπορούμε να έχουμε το παλιό σύστημα. Ναι, εντάξει, να έχουμε κάποιε αλλαγέ. Αλλά η Επιτροπή πρέπει να μα πει το, τι, τι έγινε με την παραγωγή στις χώρες εκείνες οποίες ακολουθήσαμε το ιστορικό σύστημα. Στη χώρα μου διατηρήσαμε την παραγωγή. Αυτό έγινε. Άρα λοιπόν ας μην είμαστε πολύ, α, ας μην προσπαθούμε να φύγουμε βιαστικά από το παλιό σύστημα χωρίς να αναλύσουμε ε, τα στοιχεία. Και είναι και αργά. Ε, αλλά να σας πω το εξής. Ε, τώρα, έχω, έχω ακούσει τόσο πολλού να μιλούν για την αλλαγή του ονόματο, Τι πρόβλημα έχει τουλάχιστον κρατήσουμε το C, το, το, το K, το common, το κοινή. Να βγάλουμε τη λέξη αγροτική, ε, ας αντισταθούμε. Άλλοι θέλουν να προσθέσουμε και το περιβάλλον, το θέμα των, φαγητό, των τροφίμων, εντάξει. Αλλά το βασικό ζήτημα είναι να μην ξεχνάμε σε αυτή την πολιτική το επίκεντρο, τη γεωργία και του γεωργού. Και χθε η Επιτροπή στην Επιτροπή Περιβάλλοντο, ακούσαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα καταποκοπή πληρωμών. Τι θα κάνουμε, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ποιο θα ωφεληθεί άμα συνδέσουμε το καταποκοπήν με τη γη. Α είμαστε ε, πάρα πολύ σκληροί όσον αφορά τον προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καλινόφσκι έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εδώ ε, δεν συζητάμε ε, ε, μόνο το μέλλον τη κοινή αγροτική πολιτική, αλλά το, το μέλλον του αγροτικού μοντέλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι πολύ δύσκολο να, στα πλαίσια αυτά να μην λάβουμε υπόψη τη στρατηγική 2020, μια στρατηγική που θα έχει αντίκτυπο στι προτεραιότητε για τον προπολογισμό 2000, για το, στο διαμεσονομικά πλαίσια 2014-2020. Και εδώ θέλω να πιστώ την προσοχή των συναδέλφων σε μια κάποια αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στους στόχους αυτής της στρατηγικής και στα αποτελέσματα τα οποία θα ε, προκύψουν από ε, τις ε, αλλαγές της δημοσιονομικης προοπτικής για το 2014-2020. Ο βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η αντιμετώπιση της κλιματική αλλαγής. Ναι, αλλά ο προπολογισμό μας λέει ότι θα μειωθούν οι πιστώσεις. Επομένως, η η γεωργία θα αποτελέσει αντικείμενο εκβιομηχανοποίηση το 2020. Αυτό σημαίνει ότι ε, δεκάδε χιλιάδε γεωργοί θα βρεθούν σε κατάσταση ανεργία. Και όμω στόχο στρατηγική είναι η καταπολέμηση τη ανεργία. Μια περισσότερο βιομηχανοποιημένη γεωργία θα μολύνει περισσότερο. Και όμω ο στόχο τη ε, στρατηγική 2020 είναι η προστασία του περιβάλλοντο. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι ορισμένοι θέλουν να απομακρυνθούμε από το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Ε, αργά ή γρήγορα. Μα όμω αυτό το μοντέλο μα επέτρεψε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, να προστατεύσουμε τι πολιτισμικέ αξίε, τι κοινωνικέ αξίε, την κληρονομιά μα με δύο λόγια, την κληρονομιά ε, τη κοινή αγροτική πολιτική. Κυρίε και κύριοι, ε, τώρα θα ήθελα να, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σα πω πολύ σύντομα τα εξή. Όσον αφορά την νομιμότητα τη ΚΑΠ, κατανοώ ότι όταν μιλάμε για δημόσια αγαθά, Προσπαθούμε να νομιμοποιήσουμε την ΚΑΠ και τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ. Ε, αν απομακρυνθούμε λοιπόν από αυτή τη διατύπωση, ε, τότε θα οδηγηθούμε στο τέλος της κοινή αγροτικής πολιτικής. Και όμως χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα άμεσων ενισχύσεων, ένα ισότιμο σύστημα βεβαίως. Και δεν συμφωνώ με το επιχείρημα ε, που ακούμε ότι ε, διαφορετικό βιωτικό επίπεδο, διαφορετικές πληρωμές. Ε, νομίζω ότι ε, είναι... Κοιτάξτε, όσον αφορά το βιωτικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν τόσες διαφορές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να φροντίσουμε έτσι ώστε να διατηρήσουμε κατά τα πλαίσια της ΚΑΠ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γκαρσία έχει το λόγο τώρα. Κυρία έχει ε, Ευχαριστώ, λυπάμαι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να συμφωνήσω με όλα όσα μας είπε ε, ο κύριος Μαρτίνες. Επίσης, εγώ θα ήθελα να σκεφτούμε λίγο αυτή την ΚΑΠ που μας δίνει προϊόντα μεγάλης ποιότητας, ιδιαίτερα που σέβονται ιδιαίτερα το περιβάλλον, πουθενά αλλού στον κόσμο δεν παράγονται τέτοια προϊόντα υψηλότατης ποιότητας με τόσο μικρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αλλά σε τι μας χρειάζεται κάτι τέτοιο, όταν τελικά αυτό το οποίο θέλει η Κομισιόν είναι να ξεφορτωθεί την ΚΑΠ, παρά τα καλά αποτελέσματα που μας έδωσε. Αυτή είναι η πολιτική στρατηγική των 27. Αντί δηλαδή να στοιχηματίσουν όλοι και οι Κομισιόν μαζί για αυτόν τον στρατηγικό τομέα. Πέρα από την αυτάρκεια χρειαζόμαστε ασφάλεια στην προμήθεια χρειάζεται σεβασμός του περιβάλλοντος των συμφωνιών της ΔΟΕ και προϊόντα ποιότητας και για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται και ένας κοινοτικό προϋπολογισμός. Σας ευχαριστώ και το λόγο έχει ο κύριος Γιάρ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι ε, η, κοινή αγροτική πολιτική ε, είναι καλύτερη από τη φήμη της, αν θέλετε. Λοιπόν, όλοι υπερασπιζόμαστε την ΚΑΠ Και μην ξεχνάμε ότι ε, μα προσφέρει προϊόντα άριστη ποιότητα σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε. Χρειαζόμαστε βεβαίω ένα σύστημα σταθεροποίηση των τιμών. Και ε, γιατί ε, η ποιότητα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο προστασίας. Μετά υπάρχει το θέμα της συγχρηματοδότησης. Πάντως ε, σήμερα έχουμε πολλά πράγματα κοινά, αν θέλετε. Άρα αυτά θα πρέπει να προωθήσουμε ε, στον αγώνα μας για, για την ε, προάσπιση και του προπολογισμού. Το ξαναλέω, έχουμε μια κοινή αγροτική πολιτική που είναι επιτυχημένη, μην το ξεχνάμε. Οι γεωργοί πραγματικά συμβάλλουν ιδιαίτερα στην κοινωνία και αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα σημερινά πρότυπα, αν θέλουμε να διατηρήσουμε τα σημερινά επίπεδα, τη σημερινή κοινή αγροτική πολιτική, τότε χρειαζόμαστε και τα κατάλληλα ε, δημοσιονομικά μέσα. Βεβαίω τώρα θα πρέπει να αποφύγουμε την αύξηση τη γραφειοκρατία. Αυτό θέλω να πω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπέγκερ. Danke, Herr Vorsitzender. Ich habe der Anhörung sehr ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτή την ε, ακρόαση, κυρίως ως μόνιμος ε, ε, ε, της, ε, για τον προπολογισμό, για τον πολιτή προγραμματισμό. Λοιπόν, να σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, εδώ πρέπει να δούμε τους στόχους και τα μέσα. Και θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στους στόχους και στα μέσα παρόλο που ε, σχετίζονται μεταξύ τους. Και το λέω αυτό και σε σχέση και με την πολλαπλή συμμόρφωση. Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά θα πρέπει ε, να ξεπεράσουμε και αρκετέ διαφορέ πριν μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια ομόφωνη αντίδραση του Κοινοβουλίου. Νομίζω όμω ότι η απήχηση είναι θετική γενικά σε σχέση με τον επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του περασμένου φθινοπόρου. Επρόκειτο για ένα έγγραφο τεχνικής φύσεως μεν, αλλά ε, πρέπει να καταλάβουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ότι η συζήτηση αυτή για την ΚΑΠ εντάσσεται απόλυτα μέσα σε μια ε, διαδικασία συνέχειας... δηλαδή βεβαίως και θα πρέπει να αγγλεί την έμπνευσή τη από ένα ρεαλιστικό πνεύμα, χωρίς όμως να παραμελούμε τι συγκεκριμένε ανάγκε. Άρα θα πρέπει να κατανοήσετε καλά ότι το 2012 κινδυνεύετε να βρεθείτε αντιμέτωποι με τις κυβερνήσεις σας. Γιατί, γιατί ε, οι κυβερνήσεις ε, θα, θα έχουν μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση όσον αφορά τον πολιτικό προγραμματισμό. Και θα έχω να σας πω το εξής, ότι μπορούμε να λέμε πολλές φορές όχι μέσα στην ε, ε ολομέλεια, αλλά το αποτέλεσμα που θα βγαίνει ίσως να μην είναι πάντοτε το επιθυμητό. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπέγκε. Κανιέται. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω ότι μία από τις ε, σημαντικότερες ε, πτυχές της ε, κοινωνικής πολιτικής είναι η διαφύλαξη της αξίας της πολιτικής αυτής. Και πρέπει να πείσουμε και τις άλλες επιτροπές πιστεύω ότι τα προβλήματα του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να ανταλύσουμε εις βάρος της κυρίας πολιτικής. Θα πρέπει να είμαστε θέση να έχουμε μια ΚΑΠ γερή υγιή να καλύψουμε τις μεγάλες ακόμη δυστυχώς ανισότητες μεταξύ παλαιών και νέων κρατών την απόσταση που έχουν να καλύψουν τα νεα κρατημέλη, Γιατί είναι πολύ μεγάλες διαφορές και είναι πολύ μεγάλες διαφορές βέβαια και στο επίπεδο διαβίωσης, πράγμα το οποίο δημιουργεί γενικότερα προβλήματα. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί Επίση είναι η διαφάνεια. Δεν πρέπει να έχουμε αυθαίρετα κριτήρια δηλαδή. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι δυνατόν να επαληθεύονται ε, ως προς την ευστοχία τους και ως προς την ικανοποίησή τους και ε, να είναι ε, ξεκάθαρα για τον καθένα. Μια κοινή γεωργική πολιτική δεν μπορούμε να ε, την ε, πραγματοποιήσουμε εάν δεν συζητήσουμε σε τι ωφελεί η γεωργία. Τι προσφέρει στην κοινωνία μας η γεωργία. Είναι η παραγωγή, είναι ο παραγωγός, είναι η υπηρεσία που προσφέρει στην ε, κοινωνία και πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να συζητήσουμε το ζήτημα της συγχρηματοδότησης. Με πολύ μεγάλη προσοχή υπογραμμίζω για να μην υποβαθμίσουμε την κοινωνική διάσταση αυτής της πολιτικής. Θα πρέπει να σταματήσουμε πια κάθε φορά να βρίσκουμε επιχειρήματα για την ΚΑΠ, Γιατί δεν λέμε ότι σε όλες τις χώρες τελικά οι γεωργοί είναι αυτοί που έχουν τα χαμηλότερα εισοδήματα από όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Δώσαμε ένα σωρό λεφτά στις τράπεζες για την κρίση, για το ένα για το άλλο και ποιος θα τα πληρώσει όλα αυτά. Αυτό είναι ένα βασικό σημείο στην ημερήσια διάταξη. Μετά λέμε πρέπει να φτιάξουμε ένα νέο μοντέλο. Αλλά να το θυμάστε, όχι ε, ότι, έχουμε, ότι έχει γίνει στο παρελθόν πρέπει και καλά επειδή έγινε στο παρελθόν πρέπει να το διαγράψουμε. Υπάρχουν και καλά πράγματα που έκανε η ΚΑΠ και που καλά θα έκανε να τα κρατήσουμε. Έχουμε μία νέα αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει δεν είμαστε παγκοσμίως ανταγωνιστικοί. Ε ωραία. Και λοιπόν ποιοι είναι οι όροι. για αυτόν τον ανταγωνισμό. Σύμφωνοι, ανταγωνισμός δεν υπάρχει αλλά με, με, με συγκεκριμένους όρους. Και πάμε μετά στις ε, πιο εξειδικευμένες πλευρές της ΚΑΠ. Εντάξει, έχουμε εποχιακές διαφοροποίησεις που φτάνουν μέχρι και 15% και χρειάζεται παρέμβαση στην αγορά για να μην έχουμε στρέβλωση της αγοράς. Αλλά δεν είναι οι γεωργοί που πρέπει να πληρώνουν τα σπασμένα. Και όταν μιλάμε για την ΚΑΠ, δεν πρέπει εμείς να, να θεωρούμε ότι όλα τα μέσα πρέπει να είναι τα ίδια. Πρέπει να έχουμε κατά νου την χρηματοδότηση Δεν μπορούμε εμείς να θέλουμε να γίνονται όλα αυτά ομοιόμορφα. Και γιατί να χρηματοδοτούμε άλλες πολιτικές και όχι αυτή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήταν καλό γιατί η Επιτροπή σήμερα άκουσε τη φωνή των γεωργών μας και, του κόσμου της υπαίθρου. Και θέλω τώρα να σας ε, να ε, καλωσορίσω ε, τον εκπρόσωπο από τη Βόρεια Ιρλανδία, ε, τον εκπρόσωπο των αγροτών στη συζήτηση. Είναι καλό το γεγονός ότι ακούμε ε, να ακούμε τι απόψει των Γεωργών, όχι μόνο εδώ, αλλά και στην πατρίδα μα. Πρέπει να σα πω ότι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τη συζήτηση σήμερα και πρέπει να σα πω ότι υπάρχουν ορισμένα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι ε, ξεκαθαρίστηκαν ιδιαίτερα. Ακούσαμε ε, την άποψη των Γεωργών στη συζήτηση και είναι σαφέ ότι, ότι ζητούν μια ισχυρή ΚΑΠ. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε εμεί είναι να αγωνιστούμε και στο Κοινοβούλιο και στη συνεργασία μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, να εργαστούμε λοιπόν προ το στόχο αυτό για, το, για μια μελλοντική κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013. Επίσης ακούσαμε ε, ε, ιδιαίτερα την ανάγκη σήμερα για επαρκή ε, προπολογισμό και συμφωνώ με την κυρία Μακίνες. Δεν πρέπει να δεχθούμε σε αυτό το στάδιο μικρότερο προπολογισμό. Αντίθετα θα πρέπει να ζητήσουμε το μέγιστο που μπορούμε να ζητήσουμε. Και όσον αφορά τον άλλο συνάδελφο που είπε ότι υπάρχουν στοιχεία της ΚΑΠ τα οποία ε, μας ζητούν να δράσουμε περισσότερο, ε, ίσως εδώ θα πρέπει να αναλυφθεί η δράση και από άλλα τμήματα του προπολογισμού. Πρέπει πάντως να διατηρήσουμε ένα ισχυρό σύστημα άμεσων πληρωμών και νομίζω ότι αυτό ήταν ιδιαίτερα σαφές ε, το χρειάζονται αυτό ε, οι γεωργοί. Ε, δεν το πετούν, το χρειάζονται λόγω τη κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ταυτόχρονα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη και λιγότερη γραφειοκρατία και λιγότερα εμπόδια προ τους γεωργού. Το ζητούμε να είναι πιο αποτελεσματικοί και να παρέχουν δημόσια αγαθά. Μα πρέπει να έχουν και τα απαραίτητα εργαλεία για το σκοπό αυτό. Αυτό με τη σειρά του απαιτεί συμπληρωματική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση το μέλλον της ΚΑΠ θα πρέπει να συμπεριλάβει ε, την ε, ε, κατάλληλα αγορά διαχείρισης, κατάλληλα με την αγορά έτσι ώστε να προωθήσουμε τις μακροχρόνιες επενδύσεις και να, ενισχυθούν, να ενισχυθεί τελικά το εισόδημα των αγροτών. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, να σας πω ότι η ασφάλεια, η διατροφική διακόπτει ο Πρόεδρος, η ασφάλεια, η διατροφική θα πρέπει και αυτό να, είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστώ, πάμε στο μιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συζητήσαμε όλο αυτό το απόγευμα και ευχαριστώ ιδιαίτερα στους ομιλητέ που ήρθαν εδώ και έλαβαν το λόγο. Το θέμα της κοινωνικής πολιτική πολιτικής με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ασφάλειας ε, στην αλυσίδα των ε, τροφίμων. Νομίζω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να το συζητήσουμε με τρόπο επαναστατικό, με ανοιχτό πνεύμα δεν έχουμε πλέον επαρκείς όρους για τη διαφύλαξη της ασφάλειας της αλυσίδας των τροφίμων. Πρέπει να συστήσουμε την σκοπιά του καταναλωτή. Μην ξεχνάμε ότι ο καταναλωτή είναι πολύ πιο φύλλα διακείμενος απέναντι στον ε, παραγωγό, στον γεωργό, από ότι ο ε, διανομέας, ο διανοπολιτής. Επίσης λέει ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ναι, συνεπείς πρέπει να είμαστε απέναντι στον καταναλωτή, όπως όμως πρέπει να είμαστε και απέναντι στον γεωργό όταν μειώνονται διαρκώ οι τιμέ, όταν τις εξισώνουμε τα τελευταία χρόνια συνεπώ με τις άμεσες πληρωμές, πρέπει για το μέλλον να δούμε ότι για λόγους συνέπειας δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την χρηματοδότηση, την επιδότηση. Είναι κάτι το οποίο εάν αποφασιστεί, εάν εγκαταλειφθεί δηλαδή το σύστημα των επιδοτήσεων, θα αποτελέσει μέγιστο πλήγμα για τους παραγωγούς της Ευρώπης. Επίσης, θα πρέπει πιστεύουμε ε, να συζητήσουμε τις ε, μικρότερες εκμεταλλεύσεις και το γραφειοκρατικό άχθος το οποίο έχουν να σηκώσουν, το οποίο είναι πολλές φορές δεσβάσταχτο. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε διαφορετικές ενδεχομένω λύσεις και απλούστευση των κανόνων. Ευχαριστώ πολύ. Νίκο, παρόλα. Mulțumesc, domnule președinte. Ο επόμενος Dacă nu trebuie să luăm o reducere a bugetului agriculturii ca pe un fapt împlinit... Λοιπόν, δεν θα πρέπει εμείς να δεχτούμε μυρολατρικά την ε, μείωση του προϋπολογισμού. Εμείς έχουμε την αρμοδιότητα να το αμφισβητήσουμε και πρέπει να ασκήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Στη συνέχεια, χρειαζόμαστε μεγάλη νομιμότητα. Χρειαζόμαστε μία συνενετική πολιτική, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και η αποδοχή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επίσης. Χρειάζεται επίσης αποδοχή από όλα τα κράτη-μέλη. Πρέπει να είναι λοιπόν όλα αυτά διαμφισβήτητα και ανατολικά και δυτικά. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των κρατών μελών Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις ανταγωνιστικές καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί μας. Πρέπει λοιπόν εμείς να έρθουμε εδώ με συγκεκριμένα μέτρα, να ορίσουμε ποιοι είναι οι στόχοι μας και αφού δούμε ποιοι είναι οι στόχοι μας να βρούμε τις λύσεις και τα μέσα. Λοιπόν, τελευταία τοποθέτηση και μετά ο κύριος ε, Λάιν. Ο κύριος Δανέλης έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την απόψινή διοργάνωση αυτής της ε, τόσο ενδιαφέρουσας ακρόασης και ευχαριστίες σε όλους τους ομιλητές για, την, ε, για τις πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και προβληματισμούς. Θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, πολύ σύντομα. <clears throat> Σύμφωνα με παραδοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ανακοίνωσή της για την κλιματική αλλαγή, τα κράτη-μέλη του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πληγούν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Επιπλέον όμως, αυτά θα, πληθούν, θα πληγούν και δυσανάλογα. Και αυτό διότι εκτός από αυτή καθ' αυτή την άμεση δυσμενή επίδραση, η κλιματική αλλαγή αναμένεται να πλήξει σημαντικά τόσο τις αμυγός γεωργικές δραστηριότητες, όσο και πολλές από τις εναλλακτικέ οικονομικές δραστηριότητες όπως η δασοκομεία, ο χειμερινός τουρισμός ή η εκτατική κτηνοτροφία αλλά τέτοιου είδους δραστηριότητες συχνά αποτελούν σημαντικές ή και τις μόνες πηγές διαφοροποίησης και συμπλήρωσης του γεωργικού εισοδήματος στην Ήπεθρο. Οπότε ο συνδυασμός επιβάρυνσης ορισμένων τομέων της οικονομίας και περιορισμού των δυνατοτήτων οικονομικής και κοινωνικής διαφοροποίησης στην Ήπεθρο θα είναι ιδιαίτερα δυσμενής για πάρα πολλές περιοχές του Νότου. Πόσο μάλλον που η ίδια η Επιτροπή προτείνει τη διαφοροποίηση ως τρόπο ανάπτυξης της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή, περιορισμού του ευάλωτου χαρακτήρα ορισμένων περιοχών και τελικά τον των περιφερειακών διαφορών. Ή, ακόμα περισσότερο, που περιορίζεται η δυνατότητα σε αυτές τι περιοχέ να προσφέρουν και το δημόσιο αγαθό του μετριασμού των επιπτώσεων από τι γεωρικέ δραστηριότητε. Το ερώτημα λοιπόν που απευθύνουμε μαζί με την ανησυχία μα, κυρίω αλλά όχι μονάχα προ την Επιτροπή, είναι πόσο αυτό το θέμα απασχολεί και αν ναι, τι είδους αντιμετώπιση διερευνάτε. Ευχαριστώ πολύ. Λαρία. που, αργήσαμε. Έχει και σημαντικό ρόλο στην Επιτροπή Προπολογισμού για την πολιτική. Έχει το ρόλο, Τζοβάνι. Ε, Ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο σε αυτή τη συζήτηση, γιατί εγώ πιστεύω ότι καταφέραμε να μαζέψουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία που μας χρειάζονται και για την Επιτροπή Προϋπολογισμού και για την Επιτροπή Γεωργίας. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η νέα θεματολογία για την ΚΑΠ και μέσα σε αυτούς τους νέους στόχους της ΚΑΠ θα πρέπει να παλέψουμε για να παραμείνει μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας αυτό το οποίο έχει φανεί από τη συζήτηση. είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή θα πρέπει να διατηρηθεί ο προϋπολογισμός τουλάχιστον στα επίπεδα του τωρινού. Και αν χρειαστεί θα πρέπει να προχωρήσουμε εμείς ε, για το πολιετές ε, σχέδιο για προγραμματισμού για τη Γεωργία το Κοινοβούλιο παίζει κεντρικό ρόλο στις επιτροπές του προϋπολογισμού και γι' αυτό πιστεύω η Επιτροπή Προϋπολογισμού ήδη γνωμοδοτώντας την έκθεση πρωτο, πρωτοβουλίας για το μέλλον της ΚΑΠ με εισηγητή τον κύριο Λάινων θα μπορέσει να υποστηρίξει οικονομικά μια νέα ΚΑΠ που θα επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις για τις οποίες καλούμε να απαντήσουμε. Ευχαριστώ Τζοβάνι. ο Τζορτζ Λάιον για να κλείνουμε. Λοιπόν, μη φύγετε μετά γιατί πρέπει να αποφασίσουμε κάτι. Τζορτζ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, αφού είναι και περασμένη ώρα. Ευχαριστώ καταρχά ε, του συναδέλφου για τη συμβολή του στη συζήτηση. Μα βοήθησε να διευκρινίσουμε μια σειρά ζητήματα. εμένα προσωπικώ για την έκθεσή μου ζητήματα στα οποία θα πρέπει ίσως να οξύνουμε το κείμενό μας. Εγώ θα ήθελα να σημειώσω ότι κάποτε μου είχε πει εμένα για την εκδρολογική υπόθεση που είχαμε νωρίτερα, ότι εμένα κάποιο σοφό μου είπε κάποτε ότι αν θέλω να έχω μια μικρή περιουσία, πρέπει να ξεκινήσω με μια μεγάλη περιουσία και μετά να ξοδέψω τα λεφτά στη γεωργία. Και έτσι θα καταλήξω σε μια μικρή περιουσία. Πέραν αυτού, ε, δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε τι σημαίνει η κοινή γεωργική πολιτική. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι γεωργός, είναι δραστηριότητα γεωργική, είναι δημόσιο αγαθό. Χωρίς αυτήν δεν θα υπάρχει δημόσιο αγαθό. Πρέπει, αν θέλουμε δημόσιο αγαθό, να έχουμε ικανοποιητικές συνθήκε για του γεωργού μα. Αυτό δεν μπορούμε να το λησμονούμε σε αυτή τη συζήτηση. Τρίτον, η μεταρρύθμιση για να είναι βιώσιμη θα πρέπει να είναι και ισοδική. Δεν μπορούμε να λησμονήσουμε αυτόν τον όρο. Και, τρίτο, και τελευταίον, μας το επισήμανε η κυρία Μαγκίνες. Για όνομα του Θεού, μην υποχωρήσουμε στο ζήτημα του προπολογισμού πριν καν αρχίσει μάχη. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε μια γροθιά. Πρέπει να αγωνιστούμε και όπω υπόθηκε και νωρίτερα, όταν έρθει η ώρα για την ψηφοφορία, για τι δημοσιονομικέ προοπτικέ, ξέρετε πολύ καλά ότι αν το κοινοβούλιο πει όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το λησμονήσουμε καθόλου. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και θα είναι ξέρω πολύ ενδιαφέρουσες οι επόμενες εβδομάδες και μήνες.